Proszę Państwa, otwieram posiedzenie, Κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής με το πρώτο θέμα τι έγινε στους συντονιστές θα σας πω και μετά το δύο έγκριση των σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Πριν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη θα γίνουν και ορισμένες ανακοινώσεις. Το 23 μεταφέρθηκε στον Απρίλιο το 10 η επίσκεψη στο Gateshead και το Newcastle θα συζητηθούν πριν το μεσημέρι. Πριν. περίπου στις 12 θα συζητήσουμε το θέμα των Ισπανών φαρμακοποιών και τα 11, 12 και ίσως και 15, 16, 17, 18, 19 μέχρι και 21 θα γίνουν με επισκέπτες ε, και εκπροσώπους των αναφερόντων. Πολύ δουλειά λοιπόν. Ελπίζω να μπορείτε να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Επόμενο. Τα πρακτικά της 19ης 20ης Ιανουαρίου και μετά 10 και 11 Φεβρουαρίου. Ο κύριος Ντερόσα. Η αναφορά 19 που είναι του κυρίου Γκότ έχει ένα ερωτηματικό αν θα έρθει ο αναφέρον. Το ξέρουμε ή όχι. Ο Δαβίδ μου λέει ότι θα έρθει. Ναι, αλλά δυστυχώς εγώ θα λείπω μέχρι να φτάσουμε εκεί, όταν θα φτάσουμε εκεί. αλλά μπορώ ήδη να σας πω ότι δεν εκπροσωπεί την κοινότητα που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί ο αναφέρον. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο νωρίτερα για να είμαι κι εγώ. Γιατί κατά τις τέσσερις πρέπει να φύγω. Κοιτάξτε, θα είναι ο αναφέρον εδώ ή όχι, αυτό δεν γνωρίζουμε. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσω στο σημείο 3, εγκρίση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 19ης Ιανουαρίου και συνέχεια της συνεδρίας του Φεβρουαρίου. Πριν να εγκρίνουμε τα πρακτικά, να σας πω ότι έχουμε ένα σχόλιο από τον Σε Ρόμπερτ στη συνάντηση των συντονιστών έκανε ένα σχόλιο. Είπε ότι κάποια πράγματα δεν είχαν καταγραφεί όπως υπόφηκαν. Έτσι λοιπόν υποαίρεση. Ίσως ο Σερ Ρόμπερτ μπορεί να πάρει το λόγο και να τονίσει ποια είναι αυτά τα σημεία που αμφισβητεί. Γιατί, κοιτάξτε, αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί σήμερα. Υπάρχει μια σύγκρουση σε σχέση με το τι υπόθηκε από εσά και στα πρακτικά πώς έχουν καταγραφεί. Εγώ απλώ θέλω να διορθωθούν να τα ελέγξετε και να τα διορθώσετε θέλω. Εντάξει. Εφόσον ε, θα γίνει η σύγκριση λοιπόν με τα επίσημα πρακτικά, με τα επίσημα αρχεία, θα τα εγκρίνουμε και θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά, φυσικά έχοντας λάβει υπόψη τα σχόλια του σε Πρόεδρε, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα συνεχιστεί το ζήτημα αυτό Λέμε εδώ κάτι που επιφύλαξη σε αυτή την επιτροπή. Στη συνέχεια ελέγχεται και στη συνέχεια δεν υπάρχει καμία συνέχιση. Δεν ξανακούμε ποτέ για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, ε, να πούμε ίσως ότι δεν έχουν εγκριθεί τα πρακτικά, γιατί ε, θέλουμε να ξανατεθεί αυτό το θέμα και να ξανατεθεί δηλαδή το ζήτημα αφού θα έχει γίνει ο έλεγχος, αν μπορώ να απαντήσω. Κοιτάξτε, ξέρετε ποια είναι η διαδικασία, τέθηκε το θέμα. Και αν ε, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα που να έχει να κάνει με τα πρακτικά, τότε εγκρίνονται τα πρακτικά έτσι όπως έχουν υποβληθεί. Όμως ο Σερ Ρόμπερτ είπε ότι θέλει διόρθωση των πρακτικών σε σχέση με ένα έγγραφο εργασίας ε, από δύο ομάδες εργασίας. Θέλει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα έγγραφο εργασίας, ένα working papers και ότι ήταν για συζήτηση και ξέρετε Πάντοτε πριν από το τέλος της ημέρας, αν υπάρχουν ε, διορθώσεις, δίνονται στη γραμματεία και στη συνέχεια θεωρείται ότι έχουν διορθωθεί τα πρακτικά και εγκρίνονται. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, ένα ακόμα αίτημα να μετακινήσουμε το σημείο 129 από το Β στο Α. Αυτό θα γίνει αυτόματα. Το 129 λοιπόν θέλουμε να το μετακινήσουμε από το Β στο Α και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία, ίσως στην επόμενη θητεία. Λοιπόν, οι ακόλουθες αναφορές θα πρέπει να έχουν κλείσει 7606 7987 7787 5907 και 807. Αυτό βάσει των απαντήσεων των Ισπανικών αρχών, γιατί θα έρθουν νέες πληροφορίες. 6108, 8507, 906 και 2306 θα ξανανοίξουν, γιατί έχουμε λάβει νέες πληροφορίες και καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε. Τελειώσαμε λοιπόν και με το σημείο 4, σημείο 5 διάφορα. Βάση της έκθεσης Όκεν. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλες οι αναφορές που σχετίζονται με την έκθεση αυτή θα θεωρηθούν ότι έχουν κλείσει. Ο πλήρης κατάλογος των αφορών που προτείναμε να κλείσουν θα διατεθεί στην επόμενη συνεδρίασή μας. Την επόμενη συνεδρίασή μας. Ενώ οι αναφορές που έχουν να κάνουν ε, με το δίκαιο των ακτών θα παραμείνουν ανοιχτές έτσι όπως προβλέπει το ψήφισμα. Σήμερα έχει υποβληθεί μια νέα αναφορά από την κυρία Σούζαν Βουέιτ και έχει υπογραφεί από εκατοντάδε ανθρώπους και αφορά ορισμένες καταθέσεις κατά την αγορά κίνητης περιουσίας, κάποιες προκαταβολέ όσον αφορά την αγορά κίνητης περιουσίας στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Μια ενημέρωση τη επιτροπή Αναφορών. Συναντηθήκαμε νωρίτερα με την ε, κυρία Σουσαν και λάβαμε μια αναφορά που υπέβαλε για το θέμα της νόμιμης ε, αγοράς ε, κάποιων κτηρίων στην Ισπανία και κάποιους ισχυρισμούς που έχουν να κάνουν σε σχέση με κάποιες περιοχές έξω από τη Μάλαγα. Θέλουμε να το εξετάσουμε αυτό και θα ενημερώσουμε την Επιτροπή ότι έχει κατατεθεί ε, στην ιστοσελίδα των 10 Downing Street ε, και ε, υπόψη της Βρετανικής κυβέρνησης και ξέρω ότι έχει λάβει η αναφέρουσα επιστολή εκ μέρου του Πρωθυπουργού αλλά όχι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν αργότερα σήμερα θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Το επόμενο σημείο έχει να κάνει με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Οι συντονιστές συζήτησαν δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είχε να κάνει με τη νέα διαδικασία που αφορά και τη δική μας επιτροπή Πρόκειται για τη νέα διαδικασία για τη συζήτηση στην Ολομέλεια της έκθεσης της κυρίας Όκεν. Δεν μπορούσαμε να έχουμε συζήτηση. Η κυρία Όκεν μπορούσε μόνο να κάνει μια σύντομη δήλωση και υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι και άλλες επιτροπές έχουν επιφυλάξει απέναντι σε αυτή τη νέα διαδικασία. Οι συντονιστές πρότειναν και είπα και εγώ ίδιος ως πρόεδρος αυτής της επιτροπής ότι θα πρέπει να στείλουμε μία επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, του κύριο Πέτερινγκ, προκειμένου να δηλώσουμε ότι έχουμε κάποιες αμφιβολίες απέναντι σε αυτή τη διαδικασία και από ό,τι κατανοώ και άλλες επιτροπές θα στείλουν παρόμοιες επιστολές. Βέβαια αυτό δεν θα έχει επίπτωση εργασίες αυτής της ε, κοινοβουλευτικής θητείας, κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, αλλά θέλαμε να τονίσουμε το θέμα στον κύριο Πέτερινγκ. Προφανώ können das nur unterstützen. Ich möchte aber äh, vielleicht bitten, dass man ein zweites anfügt. Προφανώς υποστηρίζω αυτό που λέτε. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να έχουμε και μια ακόμη προσθήκη. Θα ήθελα να πω ρητό στους Ιπανούς συναδέλφους ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο της έκθεσης Auken, αλλά σε άλλες επιτροπές θεωρήθηκε ιδιαίτερα δυσάρεστο το ότι πρέπει να κατατίθεται τέτοια πλήρη ψηφίσματα. Υπάρχουν πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζουν τις διάφορες αναφορές ε, και πολλές φορές μπορεί να εμπλέκονται και προσωπικά. Αλλά αν πρέπει να έχουμε τρία-τέσσερα αντιψηφίσματα, απλώ για να καλύψουμε ότι έχουμε μία μόνο τροπολογία σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αυτό είναι υπερβολικό. ακόμη και αυτοί που έχουν την καλύτερη βούληση στον κόσμο. Υπάρχει μια νέα διαδικασία με ένα πλήρες ε, αντιψήφισμα. Το υπάρχει κάτι τέτοιο όμως δεν είναι κατάλληλο, δεν είναι σκόπιμο. Και νομίζω ότι αυτό κατέστησε σαφές και με την έκθεση ΟΚΕΝ δεν υπήρχαν ε, τόσε πολλέ τροπολογίε ό,τι αφορά το κείμενο, αλλά ξαφνικά είχαμε τρία ψηφίσματα που κατατέθηκαν και πρέπει κανεί ε, να εξετάζει αν μία λέξη ένα κόμμα έχει αλλάξει κάπου. Είναι υπερβολικό αυτό, Πρόεδρο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βιλάν για την υποστηρίξη στην πρότασή μας. Ε, καταγράψαμε, καταγράψε η γραμματεία την παρατηρήσή του. Θα συμπεριληφθεί στην επιστολή που σας ανέφερα. Επίσης, να σας πω ότι συζητήσαμε εν συντομία και το θέμα της Κύπρου. Όπως γνωρίζετε ότι, εδώ και καιρό συζητάμε αυτό το θέμα και οι συντονιστές πιστεύουν ότι ίσως θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αλλά πράγματι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύθραστη η κατάσταση. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση μέχρι την επόμενη θητεία. Ο Σερόμπερτ. Ρόμπερτ. Μα είχαμε πει να μην μιλήσουμε για την ουσία του θέματος που είναι αμφιλεγόμενο και θα χρειαζόταν πολύ χρόνο, αλλά απλώς ότι έχει κλείσει η αναφορά και θέλουμε, εμείς όμως θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή μέχρι εμείς να αποφασίσουμε ότι θα κλείσει και τότε θα συζητηθούν θέματα ουσίας, όταν δηλαδή το κρίνουμε εμείς. Ο κύριος Μαυρομάτης και μετά ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Σερ Ρόμπερτ Άτκινς. Εξάλλου υπάρχει και μια επιστολή του κυρίου Δημητρίου του συναδέλφου από την Κύπρο μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία στην Κύπρο πολλών διαδικασιών. Πρώτον όσον αφορά τι ευρωεκλογέ, δεύτερον τι επαφέ που έχουν οι δύο πλευρέ και η μία και η άλλη. Κατά συνέπεια στη διαδικασία αυτή που θέλουμε και εμεί να βοηθήσουμε ω Επιτροπή Αναφορών πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η υπόθεση και η αναφορά προκειμένου να την συζητήσουμε και πάλι όπω πρέπει ανεξάρτητα το πότε. Ευχαριστώ. Tak jest. Dziękuję bardzo. Taka jest. Ναι, έτσι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν και η απόφαση των συντονιστών. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό λοιπόν και τώρα οι ψηφοφορίες... Α, ο κύριος Βίλαντ, με συγχωρείτε. Α, ναι κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ένα διαδικαστικό θέμα για την αμόχωστο. Και δεύτερον, προσθέτω κάτι σε αυτό που είχα σκοπό να πω, κάτι που με έχει ενοχλήσει πολύ. Η αναφορά για τα κέντρα νεότητος, η νεολαίας. Ζητήθηκε μελέτη, η οποία έγινε αλλά ήταν ανεπαρκέστατη όχι μόνο ως προς το περιεχόμενό της, αλλά δεν συμφωνούσε με αυτά που είχαμε αποφασίσει ως Επιτροπή. Είχαμε ζητήσει να εκταστούν τέσσερις χώρες. Δεν έγινε μελέτη πάνω σε αυτό. Και μετά έγινε κάτι, κύριε Πρόεδρε, που δεν είδα πουθενά, ούτε σε αυτήν την Επιτροπή, ούτε σε καμιά άλλη Επιτροπή. Είμαι 11 χρόνια στο Κοινοβούλιο. Ακριβώς στις 9 το πρωί ερωτήθηκε στα γλίγορα. Έχει κανένα διαφορετική άποψη και ψευτο ψηφίστηκε. Και μετά το μεσημέρι έγινε μια συνέντευξη ε, τύπου και εσείς πρόεδρο το λέω ξεκάθαρα, αυτό το οποίο κατά βάση δεν είχε αποφασιστεί. Αυτό πραγματικά είναι απαραδεκτό. Νομίζω ότι είμαι γνωστός ότι μιλάω χωρίς να λαμβάνω υπόψη ε, τα πρόσωπα ή της εθνικότητας. Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας το λέω. Γιατί σε θέματα βέβαια που μας αφορούν είμαι πάντα πολύ επιφυλεκτικός, αλλά εδώ γίνονται κάποια πολιτικά παιχνίδια στις διάφορες επιτροπές. Αλλά αυτό που έγινε εδώ με μια διαδικασία υποτίθεται είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο. Να γίνονται ψηφοφορίες, να θεωρείται επίσημη ψηφοφορία κάτι που ούτε στην ημεσία διάταξη είναι και να περνάει έτσι από την πίσω πόρτα. Να ψηφίζεται χωρίς να έχει προαναγγελθεί και να γίνεται μετά μία συνέντευξη που και να θεωρείτε ότι είναι αυτή η γενική αλήθεια και χωρίς να συμμετέχουν οι ανεφέρνε. Πραγματικά δεν έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο ε, ορίζεται στις καταστάσεις εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, ευχαριστώ όλοι οι πρόεδρος, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Τα σημείωσε η γραμματεία. και τα καταφρούν στα πρακτικά. Για αν στην επόμενη θητεία εξακολουθώ να είμαι εδώ στο σώμα και εργάζομαι σε αυτή εδώ την Επιτροπή, οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη τα σχόλιά σα. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να καλέσω τον Μάικελ να ε, διευθύνει τι ψηφοφορίε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία για την έκθεση της κυρία Γόλη για την 25η ετήσια έκθεση για την επιτηρήση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Όπως ξέρετε, θέλω στις ψηφοφορίες να είναι συνήθως κάποια ησυχία για να μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν. Ας έχουμε λίγη ησυχία και σιωπή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ουόλος. Μόλις πριν πάει τον καφέ της. Να δούμε αν έχει κανένα σχόλιο και μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όχι δεν έχω κανένα σχόλιο. Και θέλω να πιω τον καφέ μου. Ε, τώρα έφυγε βλέπετε. Um, and I the one... Και δέχομαι τη μία τροπολογία που έχει υποβληθεί. Thank you, thank you very much. There is... Ευχαριστώ πολύ. Μία τροπολογία υπάρχει. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ομόφωνα συγχαρητήρια. Κυρία Βόλης. Περνάμε τώρα στην έκθεση κυρίας Μακίνες για τη ναι, τη έκθεση σχετικά με δραστηριότητα τη Επιτροπή Αναφορών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού έτου 2008. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνη πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Θέλετε κάτι να πείτε πριν ψηφίσουμε, κυρία Όλη, ή μετά. What I'll do is give the floor to Mrs. McGuinness. Uh, if she... Κοιτάξτε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακίνες. Αν δεν το αναφέρει εκείνη θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ κυρία Μακίνες. Um, firstly, can I say... Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους τους ε, συναδέλφους που υποστήριξαν την άποψη. Δυστυχώς ο βοηθ... η αδελφός του βοηθού μου Μαρτ απέθανε σήμερα το πρωί ξαφνικά Ξέρω ότι θα θέλετε να μεταβιβάσουμε την υποστήριξή μας στον βοηθό μου και στην οικογένεια, αλλά βέβαια κατά κάποιον τρόπο είχαμε κάποια προβλήματα και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που είχα από εσά σε δύσκολου καιρού. γιατί παρόλο που πολλοί θεωρούν ότι αυτό ο τόπος είναι πολύ κρύο και γραφειοκριτό, είναι ζεστό και όλοι είμαστε μέλη μια οικογένεια. Νομίζω ο Μάρκ θα ήθελε να πει τα ίδια. Τώρα για την έκθεση θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 17 όπου δέχομαι τις συστάσεις του κυρίου Ντοράσα και της Diane Wallace και θα υποβάλω μια τροπολογία υπαριθμό 47 και ένα παράγραφο. Ίσως κατά διάρκεια της να μπορώ να παρέμβω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω το θέμα της ε, τροπολογίας εξετάστηκε, κυρία Βόλη. Εάν όχι, θα σας δώσουμε το λόγο αργότερα. Παρακαλώ, μετεβιβάστε στον Μάρκ και στην οικογένειά του τα συλληπιτήριά μου για τον θάνατο της αδελφής του. Θα περάσουμε τώρα μέσα στην πληροφορία. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 1, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 το κύριο Μαυρομάτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 Άρκιντ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω για να ελέγξουμε όμως. Ποιοι είναι υπέρ να μετρήσουμε. Υπέρ παρακαλώ. Ψηλά τα χέρια. Okay, those against. Κατά. That, that, that's carried. Ναι, εγκρίνεται, ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 6 μακίνες υπέρ.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 αναλυτικά να πούμε και όχι υπερβολικά. Υπάρχει καμιά, κανένα πρόβλημα, όχι, ωραία. Τροποποιημένη τροπολογία, 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 μακίνες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Με μια προφορική τροπολογία τερόσα. Ποια ήταν αυτή η τροπολογία. Δύο προφορικές τροπολογίες πρόεδρε. Να διαγράψουμε το τελευταίο το τμήμα της πρότασης. Και η κυρία Βάλλης θέλει κάτι να πει σχετικά με τα θύματα και την προτάσει ανακόμιση των θυμάτων. Ευχαριστώ κύριε Βόλης. Κάτι θέλετε να προσθέσετε. Ναι, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω για να ανακαταστεί αυτή η διαγραφή είναι το, η ανταπόκριση της κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον ε, Ιανουάριο του 2009 για αποζημίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σε αποζημίωση για τα θύματα. Ωραία, συμφωνείτε με τις τροπολογίες. Εντάξει, περνάμε στην τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 με 25 από κοινού. Ωραία. Όχι. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 με μια προφορική τροπολογία εντερόσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Αλλά για να μετρήσουμε ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 22 παρακαλώ. Those against. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Να ελέγξουμε και αυτό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, λάθο. Απερίφθη. Α, απερίφθη. Ναι. Άλλο σκεφτόμουν, άλλο είπα. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 28 με μάτι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 27 έχει καταπέσει. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά Αποχέ. Μάλλον είναι κρίθη για να ελέγξουμε όμως. Ποιοι είναι υπέρ της 33 παρακαλώ.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 κατά αποχές εγκρίνεται 39 έχει αποσυρθεί 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 με μια προφορική τροπολογία κύριε Μαγκίνες ναι. 43 είπατε. Για, για, για, να, για να το δω, για δώστε μου ένα λεπτό να το δω. Ο Πόντσιος μήπως θέλει... Τι ήταν αυτό. Ήθελε να προσθέσει κάτι. I Ναι, εγώ είχα αποσύρει την προηγούμενη μου τροπολογία 39 την είχα αποσύρει γιατί θεωρούσα ότι θα προστίθετο το τμήμα της ε, τροπολογίας αυτής που λέει το πρόβλημα θα μπορούσε να επιληθεί τα τη διατύπωση του παρατήματο Α σημείο 21 τη οδηγία για θέμα τη εμπορική πρακτική, αντικαθώντα συγκεκριμένα τη λέξη κατανοητή με τη λέξη στόχο τη πρακτική. Αυτό το τμήμα είναι προ 43. Ναι, είναι σωστή η διατύπωση, αλλά θέλω να είναι απόλυτα σαφέ. Παίρνουμε τη 43 με την προσθήκη του δεύτερου αυτού τμήματος 39. Ναι, μπορούμε να υποσυμφωνήσω με αυτό. Ωραία. Όπως η 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τις υπέλοιπες όλες μαζί, όχι, όχι. 46 υπέρ, κατά, Αποχές Εγκρέτη, 47 υπέρ. Η κυρία Μαγκίνες. Υπάρχει εδώ πρόεδρε μια προτινόμενη νέα παράγραφο. Θα σας τη διαβάσω. 15α. Παρατείνει η υπερβολή για απόλυτα μέλη μέρη του ψηφιασμού 550 του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη επιστροφή των περιουσιών του νόμιμου ιδιοκτήτε του στα Βερόσια. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν ορατά αποτελέσματα μέχρι το τέλο του 2008, η Αρμόδια Επιτροπή θα εξετάσει ενδεχόμενα το, να φέρει το ζήτημα των ετούντων της αμοχώς του στην Ολομέλεια. Η κυρία Παναγιωτοπούλου το έχει θυμίσει αυτό. Πρόεδρος, κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική τροπολογία. Όλοι έχουν το κείμενο αυτό. εγώ θα έλεγα να υποβληθεί σαν ε, τροπολογία για την ε, Ολομέλεια, γιατί δεν έχουν όλοι το κείμενο σε όλες τις γλώσσες. Θα ήταν νομίζω πολύ πιο δίκαιο να το κάνουμε αυτό. Διαδικαστικό, κύριο Δερόσα. Μα μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα αν έχουμε μια προφορική τροπολογία. Αντί να λέμε 2008, να πούν 2009. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα ήταν ίσως καλύτερα να μην το προσπαθούμε μετά να το τροποποιήσουμε. Το καλύτερο θα ήταν, λόγω του θέματος δεν υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, να περάσει σαν ολο... τροπολογία του στην Ολομέλεια. Ωραία. Στο επόμενο σημείο, 47 λέει ο Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ομόφωνα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. And είπατε, κυρία Μαγκίνες, να συγχαρώ εσάς, αλλά και το Μάρκ και το υπόλοιπο προσωπικό σας. Πραγματικά θα πρέπει να του φορά φόρο τιμή. Τέλο, θα ψηφίσουμε την ε, έκθεση του κ. Μαρτίνε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τροπολογίε. Επομένω, να δούμε ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο εισηγητή, κύριε Μαρτίνες. Πρόεδρε, δύο λόγια για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Θα ήθελα πάντως να είναι ενημερωμένοι συνάδελφοι για το ότι εγώ συναντήθηκα με τον Επίτροπο και εξήγησα ότι φυσικά δεν υπάρχει εχθρότητα από την πλευρά του Κοινοβουλίου απέναντι στην Κομισιόν. Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να υποστηρίξουμε τον διαμεσολαβητή και από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, δεν είναι πάντοτε μία μορφή ευχάριστη, είναι μία μορφή που απευθύνεται είτε στο Κοινοβούλιο είτε στην Κομισιόν και απευθύνει έκκληση για να επανέλθουν στην τάξη. Αλλά αν έχουμε ένα τέτοιο θεσμό, τότε καλό θα είναι να το δεκτούμε. Γιατί κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Υποθέτω πάντως ότι η Κομισιόν θα ακούσει τους δικούς μας συλλογισμούς, τους δικούς μας λόγους και ότι θα ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή μας ε, αντέδρασε όπως έπρεπε ως ένα όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν επιτρέπει να υπάρχουν εξωτερικές πιέσεις. Και πράγματι όλη η διαδικασία ήταν ε, ομόφωνη και αυτό μας δείχνει ότι είναι ισχυρό όργανο το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επιδράσει αυτό θετικά γενικά και στη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρτίνες. Ε, φυσικά θα έπρεπε να πω ότι η έκθεσή του αφορούσε τη δική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαπτής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια συνέχεια σχεδίου σύσταση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι αφορά την καταγγελία 125 καθ' 2005 ELB. Ολοκληρώθηκε τώρα η ψηφοφορία και θα ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο Λεβίσκη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Μιχαήλ Κάσμαν για την αποτελεσματικότητα του Προεδρία και ψηφοφορία. Υπάρχει εδώ η συνήθεια στις ψηφοφορίες να ζητώ να προεδρεύει ο κύριος Κάσμαν γιατί το κάνει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και τώρα κυρίες και κύριοι περνάμε στα σημεία άλυφα. Το 10 θα συζητηθεί κατά τις 12 όπως είχαμε πει και προηγουμένως. Το 11... 1249 κάθετος 2008 ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ή μήπω είναι εδώ και ο αναφέρον. Καλά. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Λέγομαι Χριστίνα Πανκόσκα και είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Μονάδα Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. αναφέρον εδώ λέει ότι είναι πολύ χαμηλή η ποιότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή North Bay της Μπάρα που είναι βορειοδυτικά της Σκοτίας, στις ε, Ευρύτες. Και ζητάει να υπάρξει ευρυζωνική σύνδεση σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές της Σκοτίας. Από ό,τι ξέρουμε, δεν έχει υπάρξει όντως ανταγωνιστική εξυπηρέτηση των ευρυζωνικών ε, συνδέσεων στην περιοχή αυτή. Και ο αναφέρον επιμένει ότι κανείς δεν ήθελε να γίνει συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές και θεωρεί ότι η λύση θα ήταν να αναβαθμιστεί να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της British Telecom και στην περιοχή αυτή στα νησιά τη Ευρύδε. Οι εθνικές αρχέ. θα έπρεπε να επενδύσουν περισσότερο στο σχέδιο ComCom παρά το ότι στη Σκοτία δεν υπάρχει. Ζητάει λοιπόν να υπάρξει παρέμβαση ώστε να δοθούν τα κονδύλια και να χορηγηθούν οι υπηρεσίες αυτές και στις ευρύδες. Η Κομισιόν λοιπόν προετοίμασε μία απάντηση και κατά αυτήν, κατά δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει όντως ασχοληθεί όπως θα έπρεπε με την ευρυζωνική σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών όπως όμως προβλεπόταν ήδη από το 2006. Ιδίω τα διαρθρωτικά ταμεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι διαθέσιμα και για τη χορήγηση ευρυζωνικής σύνδεσης στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά η αγορά δεν επενδύει καταλήλως. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εφάρμοσε ορισμένα σχέδια ευρυζωνικής σύνδεσης και στη Σκωτία και ορισμένα από αυτά συγχρηματοδοτήθηκαν εν μέρη και από τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκά ταμεία έτσι ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικοί τομείς και να μπει περισσότερος κόσμος στην αγορά εργασίας στον τομέα αυτών. Επίσης πρέπει να υπάρξει στήριξη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Δεν το αγνοούμε αυτό. Για το 2006 το ειδικό μεταβατικό πρόγραμμα η κυβέρνηση της Σκοτίας όρισε κάποια διαχειριστική αρχή και σήμερα όλα αυτά τα διαχειρίζεται το πρόγραμμα Taiwan the Taiwan. Οι συναρμόδιες αρχές λοιπόν της διαχείρισης της εφαρμογής του προγράμματος αυτού είναι αρμοδιότητά τους. Γιατί τα κράτη-μέλη αποφασίζουν εάν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα συμφωνούν ή όχι με το πρόγραμμα που έχει υποβληθεί. Το πρόγραμμά μας έχει ήδη θέσει το θέμα με τις Εθνικές Αρχές για τη Σκοτία και τον Οκτώβριο του 2008 όπου έγινε ένας πρώτος απολογισμός, η κυβέρνηση της Σκοτίας, τη ζητήσαμε από την κυβέρνηση της Σκοτίας να μας ενημερώσει για τις ευρυζωνικές συνδέσεις εκεί. Και μας είπε ότι το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό, μας έδωσε και στοιχεία αριθμητικά για τη χρηματοδότηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και είπε ότι το κόστος ή η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής συμφωνεί με εκείνη που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι αρχές του 2009 θα γίνουν και άλλες εγκαταστάσεις αλλά επίσης ότι το πρόγραμμα δεν θα ολοκληρωθεί παρά το 2011. Η Κομισιό θα συνεχίσει λοιπόν να παρακολουθεί το κατά πόσον εφαρμόζεται σωστά το πρόγραμμα και αν συμφωνεί με τους δεδηλωμένους στόχους. Αλλά το κράτος μέλος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη καταρχάς για την επιτήρηση και παρακολούθηση του προγράμματος και τη διασφάλιση του ότι η διαχείρισή του θα γίνεται σύμφωνα με τους υπόλοιπους ενωσιακούς κανόνες και με τα προγράμματα που δοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Έχω λάβει κάποιες πληροφορίες ε, ότι βρίσκεται εδώ και αναφέρον. Ε, θα ήθελα λοιπόν να του δώσω το λόγο, αλλά πριν ε, να, το κάνω αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Έχουμε λάβει πραγματικά δεκάδες επιστολές για το θέμα αυτό και ένα... Και έχουμε ένα νέο φάκελο με αντίγραφα των επιστολών από τη γραμματεία. Συγγνώμη, λέει ο μιλητής, έχουμε αντίγραφα των επιστολών που έχουν στελεί και από το Κοινοβούλιο από το House of Commons, από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νίλ Μακνέλ, ο οποίος είναι ο αναφέρον. Καλημέρα σε όλους. Λέγομαι Νίλ Μακνίλ ε, και είμαι ταχυδρόμος από την περιοχή North τη της Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συζητείτε την ε, αναφορά μου σήμερα και που μου δίνετε την ευκαιρία. Θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς ε, καταβάλαμε τις δαπάνες για να έλθουμε ως εδώ και γιατί αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο δύο είμαστε σίγουρα, μόνο δύο άτομα είμαστε εδώ σήμερα, αλλά μπορώ να σας πω ότι εκπροσωπούμε όλη την κοινότητα και οι επιστολές ε, ε, δείχνουν αυτή την εκπροσώπηση. Θα τα είχαμε στείλει με email, αλλά δεν έχουμε την κατάλληλη ε, σύνδεση. Τώρα, τα, εμάς μας αρνήθηκαν πριν τέσσερα χρόνια την ευρυζωνική σύνδεση του 2002 Δύο, οι συνδεόμενες κοινότητες ουσιαστικά πίεσε για την υιοθέτηση ενός ευρυζωνικού δικτύου. Το 2005 όμως άλλαξαν τα κριτήρια για την κάλυψη όλης της κοινότητας ε, και το βλέπουμε αυτό γιατί ακόμη δεν έχουμε ευρυζωνικές συνθέσεις. Αυτό που πέτυχαν όμως οι κοινότητες ήταν να αποκλείσουν τον North Bay και μαζί με 16 άλλες περιοχές της ε, δυτικές νήσους, ε, δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρχουν ευρυζωνικές συνδυασίε. όμως ε, πρέπει να εξετάσετε όλε τι δυνατότητε για να λάβετε τι αποφάσει. Εμεί θεωρούμε ότι έχουμε μια πολύ ακριβή ε, υπηρεσία που δεν μπορεί να εγγυηθεί την κάλυψη. Όσοι τη χρησιμοποιούν ε, όταν υπάρχει κακός καιρός ε, δεν έχουν σύνδεση και έχω γείτονες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες όταν δεν έχουμε παλήρια και οι συνδεόμενες κοινότητες το 2004 ήξεραν ότι θα είχαν προβλήματα αλλά γνώρισαν το θέμα το καιρό και communities τελικά δεν αναζήτησαν τις καλύτερες λύσεις για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Μία τοχογραφική μελέτη ε, αποφάσισε στη συνέχεια ότι θα μπορούσε να μας δοθεί αυτή η ευρυζωνική υπηρεσία, όμως η ευρυζωνική υπηρεσία σημαίνει ε, ότι ε, αν γίνεται μέσω της γης ε, πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν χρειαζόμαστε μελέτες ε, για να το επιβεβαιώσουν αυτό. Το βλέπουμε αν δεν γίνει περαιτέρω έρευνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ληφθεί μια απόφαση για το με το ποιο τρόπο θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Εμείς, να σας πω ότι κάναμε κάποια έρευνα και το περαιτέρω βήμα είναι 7,8 Έχουμε 7,8 χιλιόμετρα μακρύτερα το επόμενο σημείο σύνδεσης και ε, αν ήμασταν όμως στα 5 χιλιόμετρα μακρύτερα όλοι θα είχαμε καλύτερες υπηρεσίες για το εγγύς μέλλον δεν βλέπουμε να υπάρχει ελπίδα να έχουμε καλές υπηρεσίες, ε, αλλά εδώ περιμένουμε τέσσερα χρόνια για την παροχή υπηρεσιών και πραγματικά παράλογο εξοδεύονται αυτά τα χρήματα και ίσως να μιλάμε για ανθρώπους που να μην είναι ιδιαίτερα πολύ άριθμοι, αλλά για μας είναι σημαντική γιατί μιλάμε για τις οικογένειές μας, τους φίλους μας ε, κτλ. Για δύο χρόνια προσπαθήσαμε τους αρμόδιους φορείς στη Σκωτία να δούμε ε, πώς χορηγήθηκαν τα χρήματα και να χορηγηθούν εκ νέου για να γίνει το project. Έχουμε έχουμε γράψει περίπου χίλιες επιστολές και έχουμε στείλει πάρα πολλές αναφορές και πάλι μας αγνοούν. Το θέμα αυτό δεν είναι να έχουμε τις καλύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες, απλώς θέλουμε να δώσουμε και μία φωνή στους πολίτες, τους οποίοι έχουν αγνοηθεί από τις θεσμικές διαδικασίες. Ελπίζουμε εμείς να μπορέσετε να μας δώσετε τη φωνή μας ε, σήμερα. Πραγματικά ε, η κοινότητα αυτή χρήζει υποστήριξη και νομίζουμε, ελπίζουμε ότι θα μας τη δώσετε σήμερα. Εμείς ε, ε, βλέπουμε ότι τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης τελικά δεν συνέβαλαν στο να μας δοθούν καλύτερες υπηρεσίες το 2005. Εμεί ελπίζουμε να αναγνωριστεί αυτό το λάθος και πραγματικά να αποκατασταθούν υπηρεσίε. Δεν ζητάμε καλύτερε υπηρεσίε, ζητάμε την ίδια υπηρεσία που έχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Σα παρακαλώ, αναβαθμίστε ε, την ε, παροχή του δικτύου και σα ευχαριστώ που κάνατε αποδεκτή την αναφορά μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, να σας πω το εξή έχουμε και άλλους ακόμη πέντε αναφέροντες που θα μιλήσουν ε, πριν από το μεσημεριανό διάλειμμα. Ίσως λοιπόν να δίναμε μόνο 1,5 λεπτό σε κάθε διαφορετικά θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, δεν θα προλάβουμε. Έχουμε ακόμη δύο μιλητές, ας κλείσουμε τον κατάλογο, σας δίνω 1,5 λεπτό παρακαλώ πρώτος ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αναφέρον παρουσιάσε ε, πολύ εύγλωτα την κατάσταση. Δεν θέλω να υποστηρίζω αυτά που είπε. Ότι αυτή ήταν μια μακροπρόθεσμη εξατία Και θα έπρεπε πραγματικά οι αρχές να αλλάξουν άποψη, γιατί σύμφωνα με τις γνώσεις της τόπιας, ξέρανε οι τόποι ότι αυτό που προετοιμάζονται δεν θα ήταν εκατοποιητικό. Και θα πρέπει αυτά που είπα να τα πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Οι αναφέροντες εδώ έχουν αναφέρει τις απόψεις της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να γνωρίζει και η Επιτροπή και ο εκπρόσωπος της, Επιτροπής, της Κομισιόν ότι υπάρχει μια επιστολή όπου απαντιούνται ορισμένες ε, από τις αντιρρήσεις των αναφερόντων. Είναι επιστολή της Ιρλανδικής κυβέρνησης. ή ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής εκεί. Δυστυχώς καθυστέρησε να υποβληθεί και γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τους αναφέροντες τι φρονούν για το θέμα της κακής χρήσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης γιατί εδώ λέει ότι υπάρχει μια προσθήκη στο αρχικό σχέδιο η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο ή από τα διαρθρωτικά αλλά ότι αλλά υπάρχουν και ορισμένα σχόλια που γίνονται για αύξηση των συνδρομών στην ασύρματη, στην υπηρεσία ασύρματης σύνδεσης και δεν ξέρω τι φρονούν για όλα αυτά οι αναφέροντες. Έχει επεκταθεί όντως, έχουν επεκταθεί, έχουν αυξηθεί οι συνδρομές για την ασύρματη. Υπάρχει καμία λειτουργία που να έχει αυξηθεί ή βελτιωθεί. Ντερόσα. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως να μην έδωσα τη δέουσα προσοχή στην απάντηση της Κομισιόν. Αλλά είναι δυνατόν να απελευθερωθούν κονδύλια από την αναβάθμιση της ανταλλαγής. Σύμφωνα με την επιστολή της ε, σκοτσέσικης κυβέρνησης, ε, λένε ότι προετοιμάζεται αναβάθμιση για τις βιώσιμες ε, ανταλλαγές αν λάβουν δημόσια χρηματοδότηση έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος της ε, κυρίας επένδυσης. Είναι δυνατό κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα εδώ. Πρόεδρος. Ναι. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση για το θέμα αυτό, αλλά σας παρακαλώ μου μακρηγορήσετε, γιατί δεν μας ήταν ο χρόνος. Ευχαριστώ για το θέμα της ε, ενεργοποίησης κονδυλίων. Θα ήθελα να τονίσω το project, το έργο έτσι όπως ε, αναπτύχθηκε, χρησιμοποίησε κονδύλια από το Περιφερειακό Ταμείο και ε, έγινε μια κατανομή 4,8 εκατομμυρίων λιρών και 4,9 δόθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο και όλα αυτά δόθηκαν στο Κιούχο. Ξέρουμε ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις στα πλαίσια του project, ε, αλλά τα κονδύλια που έρχονται, με κονδύλια που έρχονται από τη σκοτσιστική κυβέρνηση είτε από την επιχείρηση. Έτσι λοιπόν το μεταβατικό μας πρόγραμμα, ως ό,τι αφορά το δικό μας μεταβατικό πρόγραμμα, νομίζω ότι αυτό δυστυχώς έχει κλείσει από χρηματοδοτική σκοπιά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι όλοι εμείς συμφωνείτε, μπορούμε να κάνουμε το εξή. Ε, θα στείλουμε μια σαφέστατη επιστολή στην κυβέρνηση της Σκοτίας, στις αρμόδιες αρχές της Σκοτίας, βάσει όσων ακούσαμε εδώ και βάσει της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήσασταν ικανοποιημένο, ε, παρακαλώ, με τέτοια εξέλιξη. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον αναφέροντα. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ε, θα θέλαμε να στείλετε αυτή την επιστολή, αλλά θέλαμε να αναφέρουμε για κάποια σημεία που η κυβέρνηση της Σκοτίας τόνισε σε μια επιστολή που έστειλε η πρωτοβουλία ευρυζωνικών υπηρεσιών δεν λειτουργεί. Υπάρχουν πολύ μεγάλα τμήματα τα οποία δεν καλύπτονται. Πολύ μεγάλα ε, τμήματα του νησιού έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα, σχεδόν το ίδιο ποσό όσο χρειάστηκε για να ε, γίνει ε, η αναβάθμιση των 370 εγκαλόγων και θέλουμε μια έρευνα να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα, θα τα αναφέρουμε στην επιστολή και φυσικά θα ζητήσουμε και τη δική σας ε, συμβουλή για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Αλλά δεν μπορούμε σήμερα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και πάλι την Κομισιόν ε, αν η Κομισιόν έχει αναλάβει έχει προβεί σε μία εξέταση στο πώς δαπανήθηκαν ε, τα χρήματα για αυτό το project ε, και θεωρεί ότι υπήρχε κάποια αξία της επένδυσης που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Κοιτάξτε, κανονικά δεν ξαναδίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δευτερολογήσει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το επιτρέψουμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει, ότι είναι ευθύνη της αρχής διαχείρισης να διασφαλίσει ότι το project από τεχνική οικονομική σκοπιά έχει παρουσιάσει τα κατάλληλα αποτελέσματα και έχει υποστεί τη σωστή διαχείριση. Επίσης, στείλαμε και εμείς πάρα πολλέ επιστολές ε, και αφού μας ε, καλέσατε και εσείς σε αυτή την επιτροπή και πάλι ρωτήσαμε την κυβέρνηση της Σκοτίας αν το project ε, παρουσίαζε τα αυτά αποτελέσματα και η απάντηση ήταν ότι τα αποτελέσματα στα οποία είχαν συμφωνηθεί ήταν ότι θα έπρεπε να λειτουργήσουν κάποιες επιχειρήσεις για να λάβουν αυτή την ευρυζωνική συνδύση και ότι αυτά τα αποτελέσματα τα είχε πετύχει το πρόγραμμα. Πρόεδρο, μάλιστα, μπορώ νομίζω τώρα να κλείσουμε τη συζήτηση και θα συνεχίσουμε όπως σα είπα προηγουμένω. Και τώρα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 12. Εδώ έχουμε αρκετές μεμονωμένες αναφορές, δεν θα τις αναφέρω, τις έχετε στην ημερησία διάταξη. Νομίζω ότι κάποιοι από τους αναφέροντες υπάρχουν εδώ στην αίθουσα. Καταρχήν ε, έχουμε την ε, Ομοσπονδία Θήρας. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μαλίτ Επιτροπής. Η αναφορά αναφέρεται σε μια δικία που θίγει τη Μάλτα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα σε πρωτοεξιακό στάδιο. Η Μάλτα είναι το πιο μικρό από όλα τα κράτη-μέλη και με τον ε, λιγότερο πληθυσμό από τα κρατη με το μόνο κράτο-μέλο ε, στο οποίο ε, η θύρα των θηρεύσιμων ειδών δεν επιτρέπεται. Εμείς δηλαδή εξαρτώμαστε μόνο από τα μεταναστευτικά φτηνά. Και λόγω αυτής της ιδιαίτερης ε, γεωγραφικής κατάστασης η Μάλτα διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο κρατός μέλος. Η Μαλτέζικη κυβέρνηση επέμεινε ε, στο να υπάρχει θύρα την άνοιξη γιατί δεν είναι διαθέσιμη κάποια άλλη ικανοποιητική λύση και η διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το σημείωσε αυτό και ποτέ δεν έφερε αντίρρηση στην πρόθεση αυτή. Η μαλτέζικη νομοθεσία σήμερα έχει μεταφέρει πλήρως στο ιστορικό δίκαιο την οδηγία περιπτυνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όλα αυτά, ε, υποστήκαμε αυτούς τους περιορισμούς, αλλά δεν επωφεληθήκαμε από τις ευκαιρίες που προσφέρει η νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε τώρα τη Μάλτα στο ΔΕΚ και αυτό καθ' αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όμως, όλα αυτά, αν ε, δούμε το ειδικό καθεστώς 77 που ε, διαπραγματεύτηκε η Κομισιόν ε, με την κυβέρνηση της Μάλτας, πιστεύουμε τώρα ότι η Κομισιόν υποσκάπτει τώρα αυτές τις διευθετήσεις, ε, γιατί μία από τις 77 διευθετήσεις που έκανε η Μάλτα με την Κομισιόν και μία από αυτές ήταν η θύρα την άνοιξη που να επιτρέπεται υπό συγκεκριμένε συνθήκες, αν αυτό τεθεί σε κίνδυνο, θεωρούμε ότι υπάρχει τάση να καταρρεύσουν και όλες οι άλλες 76 διευθετήσεις ε, που υπογράφηκαν πριν την ένταξη. Έχουμε πάνω από 31.000 υπογραφές που συλλέξαμε όχι ηλεκτρονικά αλλά από πόρτα σε πόρτα στη Μάλτα και έχουμε και άλλες υπογραφές που συλλέχθηκαν σε άλλα ε, κράτη-μέλη και οι ε, υπογραφές που συλλέχθηκαν αντικατοπτρίζουν το 10% αντιστοιχούν στο 10% του ενήλικου πληθυσμού της Μάλτα και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και τελικά εδώ μπορούμε ε, να δούμε ότι ουσιαστικά εξαπατάται ε, η Μάλτα σε σχέση με τις προενταξιακές διαδικασίες, ε, αν βλέπετε σε τι, τι υφίσταται. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Πάτρε Βέγκαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τα πρώτα σημεία. Όσον αφορά τις προελεξιακές ε, συμφωνίες, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κατά διάρκεια των συζητήσεων αυτών, για την ένταξη δηλαδή της ε, Μάλτας, εδόθη μία εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για τα πτηνά. Για να επιτρέπονται ε, η θύρα ορισμένων αποδημητικών πτηνών Άλλες εξαιρέσεις όμως δεν εδόθηκαν. Um, Malta, as is the case for all other 20... Ε, όπως τα άλλα 26 ε, κράτη-μέλη και η Μάλτα θα πρέπει να ζητήσει ειδική εξαίρεση εάν κάτι τέτοιο θέλει. Δεν υπάρχει καμία άλλη ικανοποιητική ε, απάντηση. Για τη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση η Κομισιό θεωρεί ότι η θύρα στη Μάλτα επιτρέπεται σε άλλες ε, περιόδους του χρόνου, παραδείγματος χάνει κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. βάσει των πληροφοριών που υπήρχαν, των στοιχείων για τη θύρα δηλαδή που έδωσε η ίδια η Μαλτέζικη κυβέρνηση. Γι' αυτό η Κομισιόν ε, άρχισε τον Απρίλιο του 2008 διαδικασία επιπαραβάση κατά της μαλτιατικής κυβέρνησης και το Ευρωπαϊκό Δικαστηριό θεωρήσε ότι δεν θα πρέπει να θεθεί καμία νομοθεσία από τις Μαλτεζικές αρχές ε, για την αρινή θύρα του 2009. Μέχρι στιγμή η Κομισιόν δεν έχει καμία πληροφορία ότι θα λάβει χώρα πραγματικά η αρινή θύρα το 2009. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εφαρμόζει ενιαία νομοθεσία για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση προς την Κομισιόν, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Πριν σας παρουσιάσω τις αντιδράσεις μου σε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής η Κομισιόν γνωρίζει οποιασδήποτε συμπληρωματικές συμφωνίες ή επιστολές που έχουν υπαγραφεί μέσα στα πλαίσια της ε, συνθήκης ένταξης. Ε, σημείωσα τα λόγια σας, ήταν πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν υπήρχε καμία απόκριση εκτός από κύριοι που αναφέρατε. Μέσα στα πλαίσια της ίδιας της συνθήκης. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο έγγραφο, διαφορετική δήλωση, συμφωνία. Προσωπάνα, αλλά... Σας ευχαριστώ πολύ, ελίου Θα θέλαμε να καλέσουμε την Κομισιόν να μας δώσει μια σύντομη απάντηση, παρόλο που σύμφωνα με την διαδικασία μας, η Κομισιόν θέλει να πρέπει να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Παρακαλώ, η Κομισιόν έχει το λόγο λοιπόν. Ναι, για το θέμα αυτό που δείξατε. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να δείτε ποια ήταν τα έγγραφα που υπήρχαν προενταξιακά. Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε ένα προενταξιακό έγγραφο, αλλά εγώ αναφέρομαι σε μια υπογεγραμμένη δήλωση. Όχι, δεν υπάρχει καμία συμπληρωματική δήλωση. μπορώ να σας αναφέρω αυτό το έγγραφο COM-M 110-02 του 22 Σεπτεμβρίου 2002 το οποίο έγγραφο αναφέρει ρητά ότι οι αποκλήσεις για την αερινή θύρα θα μπορέσει να εξαιρεθεί εάν αυτό χρειάζεται βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας για τα πτηνά. Czy jeszcze ktoś Μήπως κανείς άλλος ή καμία άλλη από την Επιτροπή μας θέλει να λάβει το λόγο. Α, όχι. Λοιπόν. Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Λοιπόν. Η Κομισιόν για τελευταία τελική απάντηση, γιατί δεν μπορούμε να το ζητάμε πάπυρον. Έχουν τεθεί τα ερωτήματα. Μήπως θέλετε λοιπόν να απαντήσετε στον Ευρωβουλευτή μας. Όχι, διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό. Όχι, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπα. Θέλει να δευτερολογήσει. Όχι. Δότε διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Είχα πει πριν θέσω το ερώτημα ότι θέλω να σχολιάσω μετά την απάντηση. Το είπα σαφώς ότι θέλω να σχολιάσω μετά την απάντηση για να αποσαφινιστεί το πράγμα. Αν μου το επιτρέπετε λοιπόν, πριν καταλήξει η Κομισιόν θέλω να σχολιάσω. σχολιάσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις μας είπε ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτα. Θέλετε να ξαναμιλήσετε λοιπόν. Δεν προσέχετε τι λέω. Βλέπω. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλιώς δεν θα απαντούσατε έτσι. Είχα πει ότι αποσαφήνισα ενώ μιλούσατε με τον συνάδελφό σας εκεί ότι θα σχολιάσω μετά την απάντηση της Κομισιόν. Εάν μου είχατε πει τότε ότι δεν είχα το δικαίωμα να το κάνω, δεν θα ζητούσα το λόγο. Αλλά εσείς μιλούσατε με το διπλανό σας εκεί πέρα και δεν με ακούγατε. Δεν είναι αυτός σωστός τρόπος συμπεριφοράς προς τους συναδέλφους. Και σας το λέω ειλικρινά, δεν μου φέρεστε δίκαια. Αν ακούγατε τι είπα, μιλούσατε με τον συνάδελφό σας. Δεν ακούσατε τι είπα. Πώς μπορείτε λοιπόν να με κρίνετε. Εγώ το είδα, σας έβλεπα. Σας έβλεπα. Όσο μιλούσα και τα έλεγα σαφέστατα, Είχα πει θα σχολιάσω μετά. Κοιτάξτε κύριε μου. Όχι. Κοιτάξτε δεν έχετε το λόγο. Ο αναφέρον έχει να προσθέσει τίποτα. Δεν, έχω, δεν σας πιστεύω πια κύριε Πρόεδρε και θέλω να γραφτεί στα πρακτικά, δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Την αντιπροσωπεία μας την μεταχειρίζεστε με άδικο τρόπο. Δεν είστε δικαιός. Δεν μας δίνετε την ευκαιρία να, και θα ήθελα αυτό να το αναφέρω στα πρακτικά, δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε την αναφορά μας. Διαφωνώ. Μήπως ο αναφέρον θέλει να ξαναλάβει το λόγο. Μήπως. Ευχαριστώ πράγμα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στα σχόλια του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι το εξή. Εμεί επανειλημμένω έχουμε επίσημα απευθύνει αιτήματα στην Κομισιόν ε, για να οργανώσει μια διερευνητική επιστολή επιτόπου στη Μάλτα στι ε, δύο ε, αυτές περιόδους ε, όταν δηλώνει ότι το φθινόπωρο μπορεί να γίνει εναλλακτική θύρα αντί για την άνοιξη. Ε, η οδηγία καθιστά σαφές ότι η εναλλακτική πρέπει να είναι ικανοποιητική και αυτό έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο και η Κομισιόν ποτέ δεν αξιολόγησε το τι σημαίνει ικανοποιητικός. proszę Państwa, więc myślę, że to dla Państwa... Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα και σύμφωνα με τις διαδικασίες μας θα αναμένουμε να ολοκληρωθούν διαδικασίες και στο 10. Και τώρα Κυρίες και κύριοι, ας προχωρήσουμε στο σημείο 13, αναφορά 56 καθώς 2004. Εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Κομισιόν, κυρία Σιλβία Σκατέτση, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα συνοψίσω πολύ σύντομα την υπόθεση αυτή γιατί από την τελευταία ακρόαση της Επιτροπής Αναφορών στις 26 Φεβρουαρίου 2008. Οπότε και εξηγήσαμε ποιες ήταν οι τελευταίες εξέλιξεις, δεν είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη. Επομένως, σε ό,τι αφορά την ουσία της αναφοράς αυτής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε με προσοχή. Αν οι ισχυρισμοί του αναφέροντα μπορούσαν να αποδείξουν ότι υπάρχει η παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Συγκεκριμένα ο αναφέρον υποστηρίζει ότι ορισμένα προνόμια που χορηγεί η ελληνική ομιδησία στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την ανάκτηση των δικών της ε, πιστώσεων, δηλαδή για δάνεια που δεν έχουν καταβληθεί, που δεν έχουν αποπληρωθεί, συγκεκριμένα ε, όταν έχουμε εκτελεστούς ε, τίτλους Δηλαδή όταν ε, οι συμβάσει των δανείων ε, είναι εκτελεστή τίτλη και γίνεται η αποπληρωμή μέσω της κατάσχεσης ε, των αγαθών ε, του οφηλέτη και η δυνατότητα να παρουσιάσει έφεση μόνο στο ειρηνοδικείο ο ενδιαφερόμενος ότι αυτό αντίκειται στην κοινωτική νομοθεσία. Όμως ε, θα και ότι όχι γιατί η οδηγία περί τραπεζών δεν ρυθμίζει τον τρόπο που ανακτούν τις οφειλές οι τράπεζες. Έτσι λοιπόν αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μόνη λοιπόν πτυχή που θα μπορούσε να ε, συνιστά παραβίαση της κοινωτικής νομοθεσίας είναι αυτό το προνόμιο αν ήταν τέτοιου είδους που θα αποθάρρυνε την πρόσβαση στην ελληνική αγορά άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Αλλά ούτε κάτι τέτοιο θεωρήθηκε ότι ισχύει από την Κομισιόν, γιατί Θεωρεί η Κομισιόν ότι οι τρόποι ανάκτησης μιας πολύ συγκεκριμένης πίστοσης και αναφέρομαι στην αγροτική πίστοση δεν ε, είναι τέτοιος που να αποθαρρύνει άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το να εισαχθούν και να κατασταθούν στην ελληνική αγορά. Επίσης δεν έχουμε λάβει άλλες καταγγελίες ε, από άλλες ε, ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν ε, παραπονέθηκε κανείς ότι υπάρχει τέτοια δυσκολία. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέταση της αναφοράς αυτής, ο αναφέρον επίσης έστειλε κάποιες τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ε, το ο Άριος Πάγος έκρινε αυτά τα προνόμια ε, παράνομα και αντισυνταγματικά έναντι του ελληνικού συντάγματος. Ε, και βέβαια ε, κάτι τέτοιο έχει συγκεκριμένο αντίκτυπο στο αντικείμενο της αναφοράς. Δηλαδή, αν ε, υπήρχε ούτως ή άλλως ε, κάποια παραβίαση και είχε δικαιωθεί ο αναφέροντας από το εθνικό δίκαιο, δεν θα υπήρχε νόημα γιατί να διερευνήσει η Κομισιόν. Και επιβεβαίνω ότι ακόμη και ο Εθνικός Δικαστής βρήκε συμβατία με το ελληνικό συνταγματικό νόμο και όχι με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει την ανάλυση της Κομισιόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, παραπονέθηκε ο αναφέρον ε, για το πόσο καθυστέρησε η Κομισιόν να εξετάσει την υπόθεση για να ξεκαθαρίσω ότι είχαμε δύο φορές ανταλλαγή επιστολών με τις ελληνικές αρχές. Ο αναφέρον έστειλε ε, εκατοντάδες ε, σελίδες εγγράφων που εν μέρη μεταφράστηκαν και αναλύστηκαν. Υπήρχε και νέα ανταλλαγή επιστολών ε, μεταξύ κομισιών και αναφέροντος. Έτσι λοιπόν, ε, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, εμείς θεωρούμε ότι αφού κρατήσαμε ανοιχτή την αναφορά για τρία έτη, αιτιολογήθηκε αυτό. Ήταν λογικό να τη διατηρήσουμε για τόσο καιρό. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τη δήλωση της κυρίας Ματσούκα που θα τη διαβάσουμε και ο κύριος ε, Μαυρομάρτης θα πάρει το λόγο. Η ε, κυρία Ματσούκα μας έστειλε το εξής ε, μήνυμα. Χαιρόμαστε που τα ελληνικά δικαστήρια αποφάσισαν θετικά για τον κύριο Μπαράκα σε σχέση με την Ευρω... Ελληνική Αγροτική Τράπεζα. Είναι ατυχέ όμω ότι η τράπεζα αρνείται να εφαρμόσει τι αποφάσει αυτέ. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τι επιτροπέ μα να κάνει μία έκκληση όσον αφορά την σημασία όλα τα κράτη-μέλη και συμπεριλαμβανομένες βέβαια της Ελλάδας να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να συμμορφωθούμε τις αποφάσεις που οδηγούν σε δικαιοσύνη για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρομάτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας έχει στείλει ήδη η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία και ο πρέσβης μας ε, στις Βρυξέλλες μια προσωπική επιστολή κύριε Πρόεδρε από τις 18 Σεπτεμβρίου του 2008 με την οποία δικαιώνει απόλυτα το γεγονός ότι πρώτον τα ελληνικά δικαστήρια και το ανώτατο δικαστήριο στην Ελλάδα δικαίωσε τους αναφέροντες. Όσον αφορά όμως την δεύτερη πράξη την οποία επικαλούνται οι αναφέροντες είναι ότι η Επιτροπή επί της ουσίας, η αναφορά είναι πλέον άνευ αντικειμένου εξαιτίας των ευνοϊκών αποφάσεων που έλαβε το ανώτατο ελληνικό δικαστήριο. Επίσης, όσον αφορά την Επιτροπή για την οποία ε, οι αναφέροντες μιλούν ότι αυτή ευθύνεται για κάποια θέματα όσον αφορά τη δική τους την υπόθεση, προσωπική εκτίμηση και σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή απολαμβάνει το συμπέρασμα ότι δεν έχει υπάρξει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Μιλάμε μόνο για το τμήμα που είναι το κοινοτικό δίκαιο. Για τα άλλα υπάρχει δικαίωση ήδη για τους αναφέροντες στην Ελλάδα και κατά συνέπεια η Επιτροπή δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι έχει υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαδικασία της λήψης απόφασης. Κατά συνέπεια κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει αντικείμενο πλέον όσον αφορά την δική μας επιτροπή και κατά συνέπεια οι ελληνικές αρχές έκαναν αυτό που έπρεπε. Ανώτατο δικαστήριο δικαιώθηκαν στο κομμάτι εκείνο αλλά όσον αφορά την δική μας την επιτροπή δεν υπάρχει αντικείμενο και την Κομισιόν επίσης. Ευχαριστώ. Σας Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τις προτάσεις του κυρίου Μαυρομάτη και μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Και περνάμε τώρα στο σημείο 14. Ε, αναφορά 1833-2008. Πέντε λεπτά έχει ο αναφέρον στη διάθεσή του να μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσά προσωπικά, καθώ και τη Γραμματεία τη Επιτροπή Αναφορών, όπω και τα εκλεκτά μέλη τη, τι και του κυρίου Ευρωβουλευτέ, που μα δεχτήκατε σε τόσο σύντομο μάλιστα χρονικό, χρόνο, ε, χρονικό διάστημα από την υποβολή τη αναφορά μα, προκειμένου να ακούσετε εμά του εργαζόμενου σε αυτή τη χρονική συγκυρία, στην καρδιά τη παγκόσμια οικονομική κρίση με τα γνωστά σε όλου αποτελέσματα και την άγνωση, και την άγνωση συνέχεια τη. Εκπροσωπώντα του εργαζόμενου τη Ελληνικό Χρυσό που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία τη Κασάνδρα, μπορούμε να σα διαβεβαιώσουμε ότι εμεί είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την πραγματικότητα αναφορικά με την καταγγελία. Θα μιλήσω λίγο πιο σιγά. Ε, που έχει γίνει στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και ερευνά το ενδεχόμενο παραβίασης από τις ελληνικές αρχές τη κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσει σχετικά με την πώληση των μεταλλίων της κασάντας στην εταιρεία ελληνικό χρυσό. Η έκβαση της υπόθεσης μας αφορά άμεσα, δεδομένου ότι την θεωρούμε ζωτική σημασία για εμάς και τις 2.400 οικογένειε των άμεσα και έμεσα προς το παρόν απασχολουμένων στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το δικαίωμα εκμετάλλευση των μεταλλίων τη Κασάνδρα από το 1700 έχει παραχωρηθεί στου κατοίκου τη περιοχή και από το 1893 μέχρι σήμερα σε διάφορα εταιρικά σχήματα αποτελούσε την κυρίαρχη εργοδοτική παρουσία στην περιοχή και απορροφούσε την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού. Η μεταλλευτική δράση στην περιοχή αναπτύσσεται σε μεγάλες εκτάσεις, είτε για τη λατόμευση, εξόριξη ή για την υποστήριξή τους. Οι εκτάσει αυτέ με βάση την νομοθεσία είναι δεσμευμένες αποκλειστικά για μεταλλευτική χρήση. Συνέπεια αυτού είναι για όλους τους κατοίκους της περιοχής του βορειοανατολικού τμήματος του νομού Χαλκιδικής οι δυνατότητες απασχόλησής τους να είναι συνειφασμένες κυρίαρχα, αν όχι αποκλειστικά, με τα μεταλλεία της περιοχής. <clears throat> Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 όμως, η μεταλλευτική δραστηριότητα άρχισε να εκφυλίζεται σταδιακά, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση των εργαζομένων και την αύξηση της ανεργίας σε όλη την περιοχή. Έτσι, τα τελευταία 40 χρόνια, τρία από τα εταιρικά σχήματα που είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση διαδοχικά, μετά από κάποιο χρόνο δραστηριοποίησή του, εκδήλωναν αδυναμία συνέχισή τη με αναγκαίο επακόλουθο τη διακοπή τη δραστηριότητα και τη δική μα ανεργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά σα αναφέρουμε ότι με την πάυση τη λειτουργία των μεταλλίων στι αρχέ του 2003 προκλήθηκαν μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα για τις ακόλουθες εργασίες που έπρεπε να εκτελούνται για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή, όπως ενδεικτικά οι εργασίες υποστήριξης και αερισμού των υπογείων έργων και των κεντρικών έργων προσπέλασης, ο έλεγχος και η άντληση των υπογείων υδάτων, όπως και των όξινων νερών, η ασφαλής περιβαλλοντικά απόθεση της λάσπης, από την εξουδετέρωση των νερών του μεταλλίου, η αποκατάσταση και αναβάθμιση έργων εκτροπής, η αποφόρτωση και απομάκρυνση των αδρομερών τελμάτων που περιείχαν κλπ. Σημειωτέων ότι τα κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα που προκύπτουν στα μεταλλεία και έπρεπε να γίνεται διαχείρισή, του, τους υπερβαίνουν τα 600. Το Φεβρουάριο του 2003 η εταιρεία Κίνρος, μητρική εταιρεία της TVX Ελλάς, που εκμεταλλευόταν τα μεταλλή έθεσε όλους τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα, που διήρκησε μέχρι το Μάιο του ίδιου χρόνου, οπότε και μας ανακοίνωσαν την απόφαση για πτώχευση της TVX Ελλάς, διακόπτοντας πλήρως τη μισθοδοσία των 500 εργαζομένων στα μεταλλεία. Μετά από αυτό προβήκαμε σε κατάληψη των εγκαταστάσεων και επί μήνες παραμέναμε εγκλωβισμένοι μέσα στις υπόγειες ΕΣ, στοχεύοντας την πίεση για επαναλειτουργία των μεταλλείων. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2003 έγιναν πολλές προσπάθειες να βρεθεί επενδυτής, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που θα έπρεπε ο τυχόν ενδιαφερόμενος να αναλάβει για την προστασία του περιβάλλοντος και τον αριθμό των απασχολουμένων σε συνδυασμό μάλιστα με, τον, με, άγνωστο τον χρόνο αδειοδότησης για να ξεκινήσει η μεταλλευτική δραστηριότητα. Η TVX Ελλάς το 1995 πήρε άδεια λειτουργίας για δύο μεταλλεία, εκκρεμούσε η αδειοδότησή της για το τρίτο. Στα μέσα του 2002 όμως ανακλήθηκαν οι άδειε λειτουργίας των δύο μεταλλίων και άρχισαν τα προβλήματα. Το Δεκέμβριο του 2003 έγινε η συμφωνία με την Ελληνικός Χρυσός. Το Γενάρη του 2004 ξεκίνησε η σταδιακή πρόσληψη των εργαζομένων για υποστηρικτικές εργασίες αφού δεν υπήρχε αδειοδότηση λειτουργίας των μεταλλίων. Σήμερα απασχολούνται άμεσα και έμεσα 2.400 εργαζόμενοι. Ενώ εφόσον εγκριθεί και αρχίσει να υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο που προβλέπεται στη σχετική συμφωνία, οι θέσει εργασία θα αυξηθούν σταδιακά σε 4.200 συνολικά προ όφελο των κατοίκων τη περιοχή, αν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξη. Η περιοχή μα μαστίζεται από υψηλό ποσοστό ανεργία που εγγίζει το 38% στον ανδρικό και το 42% στο γυναικείο πληθυσμό. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι για τη μεταβίβαση του ενεργητικού τη εταιρεία TVX Ελλάς στην εταιρεία ελληνικό χρυσό, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούσε να προκηρύξει διαγωνισμό εξαιτία τη πιεστικής ανάγκη να εξεύρει γρήγορα και άμεσα νέο επενδυτή, γιατί σε περίπτωση καθυστέρησης έπρεπε να απολυθεί μαζικά το προσωπικό, δηλαδή 500 εργαζόμενοι, που ήταν απλήρωτο επί 8 μήνες. Η δε πάυση τη λειτουργία της μονάδα θα προκαλούσε στο περιβάλλον τη ρήπανση που σα προανέφερα. Στι 12 Δεκάτου το ελληνικό δημόσιο, όντα επιβαρημένο με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η TVX Ελλάς το 1995 και στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πια, αφού εν ώψη των πολύ σοβαρών οικονομικών δυσκολιών τη είχε οδηγηθεί στη διαδικασία πτώχευση. Πιο γρήγορα. Ναι. Το, ε, ναι. Ε, ε, ε και λειτουργώντας εν προκειμένου με το λεγόμενο κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή βρήκε μετά από σχεδόν ένα χρόνο προσπαθειών στο πρόσωπο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Αγοραστή που θα, ανα, που θα αναλάμβανε πρώτον το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση των υπόγειων έργων, λιμνών, τελμάτων και φραγμάτων και άλλα. Δύο, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες σε επιμέρους μεταλλεία ή τμήματά τους, ώστε να γίνει δυνατή... Θα σας διαβάσω τα. Λοιπόν, από όλα αυτά που σας προανέφερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει παράνομη κρατική ενίσχυση της εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, όπως αβάσιμα προβάλλει ο ανώνυμος καταγγέλων. Οι επιλογές του ελληνικού δημοσίου ήταν αυτές που θα έκανε οποιοδήποτε ιδιώτης επενδυτή που έχει δεσμευτεί συμβατικά να διαχειρίζεται κρίσιμα εργατικά και κοινωνικά ζητήματα ή ακόμη και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Χάρη στις επιλογές αυτές του ελληνικού δημοσίου, σήμερα η ακομη και περιβαλλοντικε υποχρεωσει χαρη στι επιλογε αυτε Χρυσός σημερα η εταιρεια ελληνικο χρυσο εκτελει κανονικα τις υποχρεώσεις της για την προστασία του περιβάλλοντο και το καθεστώ των εργαζομένων, έχοντα εκπονήσει το επενδυτικό σχέδιο που έχει ήδη ε, υποβληθεί και εγκριθεί ε, επί της αρχής. Η απρόσκοπτη συνέχιση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου αποτελεί εγγύηση για τη βιωσιμότητα των μεταλλίων της Κασάνδρας και τη διασφάλιση των χιλίων και πλέον άμεσων και τριών και πλέον χιλιάδων έμεσων θέσεων εργασίας προς όφελος των κατοίκων της περιοχής που μαστίζεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε στη διάθεσή σας, όπως και η Κομισιόν, ικανά στοιχεία για την υπόθεση και ζητούμε μαζί με τα σεβαστά μέλη της Επιτροπής σας να δοθεί το δυνατόν συντομότερο θετική λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει αφού για μας και τις οικογένειές μας αποτελεί θέμα επιβίωσης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Dziękuję bardzo. Przedstawiciel Komisji, pan Dimitrios Pikios. Bardzo proszę, Παρακαλώ, κύριο Σπίκη, παρακαλώ να είστε euh, Λέγομαι Μέλιο Σινγκ. Θα είμαι κατά τα δαρατών σύντομο. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι πράγματι ε, η Κομισιόν άνοιξε μια διαδικασία σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την πώληση για 11 εκατομμύρια στην ε, εταιρεία Ελληνικός Χρυσός των λόγο λόγω ορυχείων. Κάναμε μια προσφυγή. Μια που αυτή η πώληση έγινε χωρίς να ανοίξει διαδικασία υποβολής προσφορών και σας λέω ότι η Κομισιόν είχε αμφιβολία στον αφορά την τιμή που κατεβλήθη από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός για την αγορά των ορυχείων αυτών. Και ο στόχος διαδικασίας που ξεκίνησε πέρσι το Δεκέμβριο η Κομισιόν ήταν ακριβώς να επιβεβαιώσει κατά πόσον η τιμή που κατεβλήθη ήταν τιμή αγοράς. Ε, αυτή τη στιγμή δημοσιάσαμε την ε, έναρξη της διαδικασίας στην επίσημη εφημερίδα. Τα ενδιαφερόμενα μέλη εκλήθησαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αναλύει τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και δεν μπορώ παρά να καλέσω να αναφέρω αν έχει καινούργια στοιχεία να τα μεταβάσει το γλυκορότερο δυνατό στην Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η Κομισιόν δεν πήρε οριστική απόφαση. Θα το κάνει υπό το φως όλων των σχολείων που θα λάβει. Και φυσικά δεν υπάρχει εκ των προτέρων θετική ή αρνητική στάση. Υπάρχει μια φυσιολογική διαδικασία σε κάθε τέτοια περίπτωση ανίζει αυτή την διαδικασία η Κομισιόν. Ο κ. έχει το λόγο. Παίρνω το λόγο σήμερα γιατί όπως ακούσατε από τους αναφέροντες υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα οικονομικό, οικονομικής κρίσης, ανεργίας και όχι μόνο στην περιοχή αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ στεκόμαστε όμως σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου από το 1600, 1600 είναι η περιοχή ακριβώς που ασχολείται με αυτό το θέμα φτάσαμε σήμερα σε ένα σημείο τέτοιας κρίσης που η Επιτροπή λέει ότι προχωράει στα θέματα για τα δημοσιεύματα και τα λοιπά στην εφημερίδα, της, ε, στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χωρίς όμως να εξετάσει και μια λεπτομέρεια την οποία δεν άκουσα την Κομισιόν. Ζητούσε, ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να καταθέσει ένα στοιχείο το οποίο στοιχείο σήμερα έχει ήδη περιέλθει και το έχω και εγώ και το οποίο δεν άκουσα. Είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει αυτά τα οποία έχει ζητήσει η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, όταν εδώ δικαιολογημένα και με αριθμούς του οποίου ζήτησε η ίδια η Κομισιόν αναφέρεται ότι είναι νόμιμα και όχι παράνομα και δεν υπήρχε, έχει υπάρξει τέτοια χρηματοδότηση που αναφέρονται, το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να προχωρήσουμε για να δώσουμε θέσεις εργασίας προστασία του περιβάλλοντος από έναν αναφέροντα. Και πολύ σωστά εδώ με ευγενικό τρόπο είπαν οι αναφέροντες ότι σαφώς ένας αναφέρον ανώνυμος, δεν θέλουμε να τον αναφέρουμε, έκανε αυτή την αναφορά. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι αυτή μετά την τελευταία πλέον επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης του ελληνικού κράτους αυτό το θέμα δεν μπορεί να έχει συνέχεια από την Επιτροπή. Η γνώμη μου λοιπόν είναι για να μην μείνουν οι εργάτες απλήρωτοι όπως έχουν μείνει και χωρίς δουλειά σε αυτή την κρίση προσφέρεται μια εταιρεία να δώσει εργασία. Δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα ως Επιτροπή Αναφορών και γεγονός είναι ότι η Κομισιόν δεν μπορεί πλέον να κρατήσει ανοιχτή αυτή την υπόθεση διότι πήρε τα στοιχεία τα οποία σαφώς έχει και στα χέρια της και τα οποία σήμερα δεν ακούστηκαν εδώ. Ευχαριστώ. Carlos presidente. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ακούσαμε την Κομισιόν και το ακούσαμε όλοι σε αυτή την Επιτροπή. Αν η Κομισιόν δεν έχει καταλήξει ακόμη σε μια θέση ούτε υπέρ ούτε κατά, εγώ πραγματικά εμπιστεύομαι τα όσα είπε ο κύριος Μαυρομάτης και με τα έγγραφα που παρουσιάζει και με τα σχόλια που κάνει, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε την ε, αναφορά αυτή, Πρόεδρε. Πρόεδρος, θα ήθελα να αναφερθώ στους συντάκτες της αναφοράς. Ακούσατε, να απευθυνθώ στους συντάκτες της αναφοράς. Ακούσατε μόλις τι μας είπε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι περιμένει περαιτέρω πληροφορίες και δεδομένα και ακούσατε και τον κύριο Μαυρομάτη ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει κατά την αποψή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα πρέπει να κλείσει το θέμα. Και ο κύριος Καρλός Τουρκές πιστεύει ότι θα πρέπει να κλείσει η αναφορά. Θα ήθελα εσείς να λάβετε μια θέση κατόπιν όλων όσων ακούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε παρακαλώ να τοποθετηθείτε. Ναι, το μόνο που θα ήθελα και εγώ να αναφέρω εκ μέρους όλων των εργαζομένων της ε, Ελληνικός Χρυσός είναι ότι και εμεί συμφωνούμε με την τοποθέτηση του κυρίου Μαυρομάτη ότι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να κλείσει αυτή η υπόθεση, γιατί φοβόμαστε ότι αν δεν κλείσει θα δημιουργηθούν προβλήματα πολλά ξανά για μια πολλωστή φορά για εμά και τι οικογένειε μα εκεί πάνω. Και ίσω και μια συμπλήρωση να κάνω, ε, το περιβαλλοντικό θέμα που υποτίθεται ότι αφορά τον καταγγέλλοντα δεν αφορά μόνο αυτόν, ενδιαφέρει και εμά, γιατί εμεί ζούμε εκεί, Αυτό ο καταγγέλλοντα δεν ξέρουμε που, ζουν, που ζει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να αναφέρω, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ακούσατε και εύχομαι να, να λήξει θετικά για όλους μας αυτή η υπόθεση. Καλά, αφού όλοι συμφωνούν να κλείσει η υπόθεση, να την κλείσουμε την αναφορά. Κύριε Μαυρομάτη. Κρίνω και δεν θέλω να κλείσει η αναφορά σαν να μην υπάρχει είναι ότι το θέμα της Κομισιόν δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης για συνέχεια. Αυτό όλο το θέμα είναι με αυτό που κατέθεσα ήδη τα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης που κατατέθηκαν όπως ζητήθηκαν από την Κομισιόν και ποια δικαιολογεί απόλυτα αυτό το θέμα. Άρα η αναφορά μπορεί να μείνει ανοιχτή για την δική μας την Επιτροπή δεν σημαίνει όμως ότι το θέμα όλο από την πλευρά της ε, Κομισιόν πρέπει να μείνει ανοιχτό, πρέπει να κλείσει από την Κομισιόν όλη η υπόθεση. Τότε λοιπόν, αφού ο κύριο Μαυρομάτης μας διευκρίνησε ποια είναι η άποψή του, τότε εμείς θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Please sit down everybody, because... Καθίστε παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Yes, yes, but...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 το επόμενο θέμα μας είναι το 15 αναφορά 1248 κάθετος 2007 του κυρίου Ραφάλ Γκαβρόνσκι. Μήπως είναι παρόν, είναι. Έχει λοιπόν το λόγο για πέντε ολόκληρα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, σας κατευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω την αναφορά μου. Είναι η δεύτερη σχετική αναφορά. Η πρώτη είχε θεωρηθεί απαράδεκτη. Και ο συναναφέρον είναι εκείνος που είχε καταθέσει την πρώτη. Είχε πει τότε ότι ότι ή θα αυτοπυρποληθεί ή άλλος θα αυτοκτονήσει άμα δεν λήξει το θέμα του. Και μάλιστα μπροστά στην Πολωνική Βουλή. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των εκτροφέων αλόγων της Πολωνίας και το θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σχετίζεται, σχετίζεται λέγω, με την επιστροφή των κτημάτων που παράνομα είχαν κατασχέσει οι άνομοι κομμουνιστές. Εγώ δεν πήρα παρά μόνο μερικές αποζημιώσεις και όχι όσες έπρεπε, αν και ε, είχα συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την οργανική γεωργία, για τη βιολογική γεωργία και φυλακίστηκα και για τέσσερις μήνες αφού επισκέφθηκα και το Στρασβούργο και γι' αυτό θεωρώ ότι με δίωξη και εγώ και τα άλλα μέλη της μη κυβερνητική οργάνωσής μας. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα δύο πτυχές του προβλήματος. Η ιδιοκτησία, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι προβληματικό γιατί μπορεί κάποιος να διωχθεί πολλές φορές για το ίδιο αδίκημα. Και αυτό λέει το ποινικό δίκαιο στην Πολωνία το επιτρέπει. Στην περίπτωση μας δε δεν έχω τη δυνατότητα να, να μετανοήσω για την παρανομία μου γιατί ο νόμος σε άλλες χώρες προβλέπει τη δυνατότητα συμφιλίωσης μηνύοντος και μηνυτού, αλλά στην Πολωνία όχι. Πώς να πληρώσω το έγκλημά μου λοιπόν. Ο πρόεδρος σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποιο είναι το πρόβλημα που θέτει η αναφορά. Εμείς ε, για να σας βοηθήσουμε είμαστε εδώ, αλλά πια ξεκαθαρίστε το μας θέλω τις αποζημιώσεις μου γιατί είμαι βιολογικός καλλιεργητής και οι επιθεωρήσεις που έγιναν τέσσερις φορές είχαν θετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερον, η παραβίαση του άρθρου 6 της συνθήκης της Ένωσης. Ιδιαίτερα δε παράγραφοι 1 και 2 Παραβίαση από την πολωνική κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τους κανόνες μας, αφού μίλησε ο αναφέρον, τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και μετά θα συζητήσουμε. Ο κ. Ιστβαν Βάγε. από την Κομισιόν. Πρόεδρε. Λέγομαι στον Βαράρειας. Εργάζομαι στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Ανάπτυξη της Υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, διάβασα προσεκτικά την αναφορά σας και να σας ενημερώσω καταρχήν για το, το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προβλέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει αρμοδιότητα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με ποινικέ έρευνες, με ποινικέ διαδικασίε στα κράτη-μέλη. Ούτε έχουμε αρμοδιότητα να διασφαλίσουμε την προστασία της οικογένειάς σας. ή να ρυθμίσουμε, παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουμε διάφορους ισχυρισμούς που προέρχονται από ολοκληρωτικούς θεσμούς που εξακολουθούν να υπαρχούν στην Πολωνία. Πάντως, έχω εκφράσει την απόψή μου για τη δική σας υπόθεση. Όταν ε, ζητήσατε άμεση ενίσχυση, Αυτό είναι ένα θέμα αρμοδιότητας κοινοτική. Καταρχήν, να σας πω πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των ταμείων. Εσείς τελικά ζητήσατε χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Αλλά με τα κράτη-μέλη έχουμε κοινή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη γεωργία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση αυτών των αιτήσεων γίνεται από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την ευθύνη να αναθεωρεί το συνολικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο ε, της εκαθάρισης των λογιστικών διαδικασιών. Αυτό το πράξαμε και στην περίπτωση της Πολωνίας και από ό,τι καταλαβαίνω στην καταγγελία σας ε, αναφέρεστε σε κάτι που έγινε το 2004. οι έλεγχοι που θα γίνουν, ε, ε, η διαχείριση των οκτώ καταγγελιών και η έγκριση των πληρωμών, όλα αυτά τα αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης. Επομένως, μόνο τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα να αποφασίσουν επί μεμονωμένων περιπτώσεων, όπως είναι η δική σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, δεν εμπλέκεται κατά αυτόν τον τρόπο στην ε, γενική αναθεώρηση. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένες υποθέσεις, φυσικά η απόφαση λαμβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε έφεση κατά των αποφάσεων των εθνικής διοίκησης, να προσφύγεται στο δικαστήριο και το πολωνικό δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έτσι όπως εφαρμόζεται, σε σύγκριση και με το πώς εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είμαι έτοιμος να απαντήσω τις ερωτήσεις σας σε σχέση με τις ε, συνθήκες, με τους όρους επιλεξιμότητας. Αν ε, θέλετε να ξέρετε πώς ορίζουμε το γεργό κτλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει ότι η Κομισιόν δεν ε, είναι επαρκώ αρμόδια για να παρέμβει σε μια τέτοια υπόθεση, αλλά η δική μα Επιτροπή έχει ευρύτερε αρμοδιότητε. Και θέλω να σα πενθυμίσω ότι όταν ε, μιλάμε για άδικη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Πολωνία, σε συγκεκριμένε περιπτώσει, τότε η δική μα Επιτροπή υπενθύμησε στις εθνικές αρχές ποιες είναι οι δικές τους ευθύνες και οι τοπικές αρχές ε, έδρασαν κατάλληλα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον αναφέροντα και θα ήθελα πραγματικά να παρουσιάσετε την ουσία της υπόθεσης και ίσως μπορείτε να μας παρουσιάσετε και τις δικές σας προτάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τον αναφέροντα σε κάποιον ε, άλλο κύριο θα δώσω το λόγο, γιατί εσείς είστε δικηγόρος, λέει ο πρόεδρος, και θα ήθελα να, κύριε και να πάρετε το λόγο και να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον αναφέροντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά και μου δίνετε και το λόγο. Εγώ είμαι μέλος μιας άλλης επιτροπής, δεν με ξέρετε. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Γεωργίας και ε, ασχολήθηκα με το θέμα του κ. Καφρός στην Πολωνία όταν μου το είχε παρουσιάσει. Νομίζω ότι βέβαια το θέμα των αμέσων πληρωμών είναι σημαντικό. Μπορεί όμως να επιληθεί σε επαφέ με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η υπόθεση του κυρίου Γκαβρόσκη είναι πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή. Όχι επειδή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στην απόφαση του δικαστηρίου. το δικαστήρια είναι ανεξάρτητα προφανώ. Αλλά το θέο είναι κατά η διπλή δίωξη, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι γεωργό και καταρχήν κατηγορήθηκε ότι πήρε κάποια χρήματα άδικα, αχρέωσα. Και τιμωρήθηκε διπλά. Καταρχήν του αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, πολύ σημαντικό ποσό, Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη ήταν ε, ότι κατηγορήθηκε με το να έχει εισπράξει τα χρήματα αυτά εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατηγορία. Στην επίσημο κατάλογο δηλαδή των κατηγοριών αναφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα από τα θύματα των ε, πράξεων του κυρίου Καβρόσκη σε ποινικές διαδικασίες αυτού του τύπου, οποιοδήποτε θεωρείται ότι ή ε, έχει κάνει κάποιο έγκλημα, έχει το δικαίωμα να συναντήσει το θύμα και να προσπαθήσει να βρει μια λύση. Ίσως ο κατηγορούμενος δεν, δεν θεωρείται πια υπεύθυνος, ίσως ε, η, η τιμωρία ήταν πάρα πολύ βαριά. Εδώ ένα από τα θύματα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα θέλαμε στο δικαστήριο στην Πολωνία να υπάρχει κάποιος πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μιλήσει ως θύμα. Βέβαια το δικαστήριο στην Πολωνία δεν ήξερε ακριβώ τι να κάνει. Κάποια στιγμή Είχα και εγώ εμπλακεί στο θέμα της λειτουργίας των δικαστηρίων ε, στην Πολωνία και ξέρω ότι συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν σωστή η απόφαση που ελήφθη. Εκρατήθη για τέσσερις μήνες στην Πολωνία ο κ. Γκαβράουσκι. Αυτή είναι πολύ εξαιρετική κατάσταση. Μίλησα σε διάφορους συναδέλφους για το θέμα αυτό. Μου συναδέλφους από διάφορα κράτη-μέλη. Και μέχρι στιγμή κανένα δεν είχε ακούσει μια παρόμοια υπόθεση. Με υπόθεση κατά την οποία ένα γεωργό και δεν είναι η μόνη η περίπτωση του κ. Γκαβρόσκη αυτού του τύπου στην Πολωνία, όπου λέει ένας γεωργός κατηγορείται ότι πήρε τα χρήματα αχρεωστήτως και γι' αυτό το λόγο φυλακείται. Για πιστεύουμε ότι αυτή η περίπτωση, η περίπτωση του κ. Γκαβρόσκη, που φυσικά εσείς κύριε Πρόεδρε θα λύσετε το θέμα του τι πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον όμω πρέπει να στείλουμε μια επιστολή προς την πολωνική κυβέρνηση ώστε και που να λέει ότι αυτές, αυτό το πρόβλημα πρέπει να θεωρηθεί ότι ακολουθεί ειδική διαδικασία, δηλαδή ότι το παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η προστασία, για να το πω έτσι, Νομίζω θα βοηθήσει τον κύριο Καβρόνσκι. Ξέρω ότι τέτοια μέθοδος έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν, υπάρχει προηγούμενο και δεν θα αποτελεί παραβίαση των προβλεπωμένων από την Πολωνία, να μας τα εσωτερικά της κλπ. Τέλος, το θέμα της διπλής δίωξης για το ίδιο παράπτωμα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να στείλετε επίσης μια σχετική επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση και στην Κομισιόν ταυτόχρονα, ώστε όπου να ζητάτε να πάυσει πια αυτή η υπερβολική δίωξη και η επιβολή προστήμων αφού έχει επιβληθεί πρόστιμο, δεν χρειάζεται και ποινική κύρωση, γιατί εδώ είναι δύο φορές διπλή τιμωρία για το ίδιο παράπτωμα. Για αυτή την περίπτωση αρκούν αυτά. Αλλά πιστεύω ότι εσείς τώρα θα δείτε ως Επιτροπή Αναφορών αν θέλετε να γράψετε την επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση που σας ανέφερα. Το σημαντικότερο θέμα όμως που τίθεται είναι εδώ η διπλή δίωξη. καθώς και η παρακολούθηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι καινούριο στις ποινικέ διαδικασίες της Πολωνίας, γιατί μέχρι τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση την... Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απούσα σε τέτοιου είδους ποινικέ διαδικασίες. Τώρα μπορεί να πρέπει να απευθυνθείτε στην νομική επιτροπή ή στην νομική υπηρεσία σας. Ένα λοιπόν να γράψετε επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση ώστε να παρακολουθηθεί η υπόθεση και δεύτερον και η πολωνική κυβέρνηση και η Κομισιόν να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα της διπλής διώξης. Ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν το εξής. Θα στείλουμε επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση, όχι στο δικαστήριο βέβαια, στην κυβέρνηση, στις πολωνικές αρχές και μας είπατε επίσης και προς την Κομισιόν για το θέμα της και, για τα δύο θέματα. Πρώτον, την εκπροσώπηση της Ένωσης στην παρακολούθηση δικών τέτοιου είδους και δεύτερον στη διπλή δίωξη. Θα δούμε λοιπόν το περιεχόμενο των γραμμάτων, θα το δείτε ίσως και εσείς και μετά θα τα στείλουμε. Αμέσως μετά από τη συνεδρίαση ή αύριο θα ζητήσουμε από τη γραμματεία να διατυπώσει καταλήλω τα δύο γράμματα προς την πολωνική κυβέρνηση και προς την επιταροπή συγκομισιών. Αυτά για σήμερα. Θα σας τηρούμε ενήμερο. Και τώρα το επόμενο σημείο. Σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει από την αρχή, πρέπει να επανέλθουμε σε ένα σημείο για το οποίο δεν έχουμε πολύ χρόνο, το 10. Το 10. Η επίσκεψη στο Gateshead και Newcastle. Five minutes, yes, thank please, you, maximum, or, or less. Or thank you very rather much. less. Πέντε λεπτά, πέντε λεπτά maximum, ε, πέντε λεπτά. Μα θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων και εγώ και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί του Gatehead για την επίσκεψη και εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους ήκουσε ενώ οι εθνικές αρχές δεν τους ήκουγαν. Και αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει άμεση, μπορεί να υπάρχουν άμεσες επαφές μεταξύ λαού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναφορά που έγινε η έκθεση για την επίσκεψη είναι κάτι που το δέχομαι και θα ήθελα να προτείνω ότι ένα σημείο της μπορεί να ενδυναμωθεί στις συστάσεις στο σημείο 2 λέει ότι τα περιβαλλοντολογικά πρέπει να υπάρχουν μόλις το αέρα και επιστημονική παρακολούθηση αλλά ένα από τα προβλήματα που είδαμε εκεί είναι ότι τα υπόγεια ύδατα ή τα επίγεια, τα επίγεια μάλλον ύδατα, πρέπει να παρακολουθηθούν ιδιαίτερα γιατί οι επιπτώσεις μιας μόλυνσής τους θα ήταν τεράστιες. Μετά την επίσκεψη, στα τέλη Φεβρουαρίου, υποβλήθηκε νέα έκθεση για αξιολόγηση των υδροχεολογικών κινδύνων. Και εκεί αναφερόνταν και τα επίγεια ύδατα. Άμα θέλετε μπορώ να σας δώσω αντίγραφο πριν για να δείτε μήπως χρειάζεται να το λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Καλά. Νομίζω ότι θα τα λάβουμε υπόψη μας αυτά που είπατε και θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία αφού μας υποβάλλετε το έγγραφο που είπατε. Και τώρα κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε με το 16. Είναι ολόκληρη σειρά αναφορών για τους Ισπανούς φαρμακοποιούς. Οι αναφέροντες είναι πολλοί, αλλά επειδή πρέπει σε 20 λεπτά να τελειώσουμε, ερωτώ πόσοι θέλουν να λάβουν το λόγο από εσά, πόσοι. Έχω έναν αρχικό κατάλογο, αλλά βλέπω ότι 7 θέλουν να λάβουν το λόγο και άρα 2 λεπτά ο καθής και η καθεμία. Κύριο Χαβιέρ Πιμενικράου. Δύο με δυόμιση λεπτά και μετά ο Μαρτίνες Ρέι, Πέρες και Μοράλες. Αλλά δύο λεπτά ο καθένας και η καθεμία. Ο κύριος Χαβιέρ Κράου πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση εδώ. Ε, το Σώμα της Βαλένσια ζητά να θέσει τέλος το Κοινοβούλιο στη διαδικασία υπερβάση κατά της Ισπανικής οποθεσίας ε, για τα φαρμακεία και να ξεκινήσει μια κοινοβουλευτική συζήτηση ε, όπου θα εξετάζεται το σύνολο του τομέα και θα συμμετέχουν και άμεση εκπρόσωποι, ευρωβουλευτές, πολίτες και ενώσεις. Φαίνεται ε, ότι η Κομισιόν ε, ουσιαστικά ταυτοποιεί το σύστημα της απελευθέρωσης ότι είναι το τέλειο σύστημα για όλα τα κράτη και κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να το επιβάλλει μέσω της διαδικασίας επί παραβάση. Αυτό ουσιαστικά δεν συνάδει με το δόγμα του ίδιου του Ευρωκοινοβουλίου. Όταν το Κοινοβούλιο μελέτησε την οδηγία για τις υπηρεσίες, απέκλεισε τις υγειονομικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τις φαρμακολογικές υπηρεσίες από την απελευθέρωση της ε, χορήγησης της παροχής υπηρεσιών. Επίσης, ε, θα ε, αντίκειτο αυτό σε άλλες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Ένωση, σύμφωνα με τις οποίες δεν πρέπει να έρχουμε εναρμόνιση οι διαδικασίες απελευθέρωσης σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλες οικονομικές δομές, αλυσίδες, μεγάλα εμπορικά φαρμακεία που θα εισαχθούν ε, στην Ισπανία και ε, αυτό με τα ανάλογα αποτελέσματα. Έχουμε κάνει και διάφορες μελέτες και σε μία μελέτη έχουμε μελετήσει την εγκατάσταση των φαρμακείων σε όλη την Ευρώπη και από τη μελέτη αυτή μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι στις χώρες όπου υπάρχει απελευθερωμένο σύστημα φαρμακείων την ιδιοκτήτη ιδιοκτησία ε, των οποίων ε, ε, την έχουν επιχειρήσει. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε φαρμακεία που είναι πολύ πιο μακριά από τον πληθυσμό. Ενώ στην Ισπανία το 99% του πληθυσμού έχει την εγγύηση, ακόμη και οι τουρίστες, δηλαδή αυτοί που έρχονται στη χώρα μας σε ορισμένε περιπτώσει, περιστάσει, συγγνώμη, όλοι μέσα σε πέντε λεπτά να μπορούν να μεταβούν στο φαρμακείο και να αγοράσουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλε χώρε, όπου η απελευθέρωση έχει οδηγήσει στο να έχουμε φαρμακεία πολλά χιλιόμετρα μακριά από όπου ζουν οι ηλικιωμένοι και ασθενείς. Έτσι λοιπόν ζητούμε από την Κομισιόν να σταματήσει τη διαδικασία επί παραβάση και να ξεκινήσει τη συζήτηση προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού πολίτη σε ό,τι αφορά της, ε, την ε, παροχή φαρμακολογικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέη, δύο λεπτά. Εγώ εκπροσωπώ την Ένωση Καταναλωτών στην Ισπανία. Ε, Έχω να πω ότι βλέπουμε να γίνονται αλλαγέ σε μια ισχυούσα αγορά και δεν θα υπάρχουν καμιά φορά αρνητικέ επιπτώσει. Από την άλλη μεριά όμω εδώ δεν έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί στην Ισπανία με επιτήρηση των ε, εθνικών αρχών και οι φαρμακοποία αυτοί χαιρούν της εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ε, οι καταναλωτές χρειάζονται ελευθερία επιλογή. Εμείς προσπαθούμε να δούμε ποιος κερδίζει από την αλληλεγγύη αυτή. Ίσως οι μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μετά που θα έχουν φτάσει οι τιμές σε ένα επίπεδο σταθερότητας και οι μικρές επιχειρήσεις θα απορροφθούν από τις μεγάλες αυτές ή θα φτωχεύσουν. Δεν θα ωφεληθεί καθόλου δηλαδή ο καταναλωτής από την απελευθέρωση αυτή των υπηρεσιών. Ε, ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε απομακρυνθεί πολύ από ένα κρατικό μονοπολιστικό σύστημα. Έχουμε περάσει ένα ιδιωτικό μονοπολιστικό σύστημα. Η προτίμησή μας είναι να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, να είναι κοντά εκεί που μένουν οι καταναλωτές, να μην χρειαστεί να πάνε σε κάποια μεγάλα κέντρα ε, εμπορικά ο πληθυσμός ε, γεράσκει, πολλοί δεν οδηγούν αυτοκίνητο. Πώς θα πάνε να βρουν τα φράματά τους οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα σφάλματα άλλων. Σας ευχαριστώ. Ντολόρες που τρία με λεπτά. Como representante ως ε, εκπρόσωπος ε, της Ένωσης ε, Αρθρίτιδας της Βαλένσια. Εγώ υπερασπίζω το μεσογειακό μοντέλο για τους εξής λόγους. Ή όσοι έχουν αρθρίτιδα και άλλοι ασθενείς πάσχουν από μία χρόνια ασθένεια, έχουν δυσκολίες πρόσβασης για να αναζητήσουν τα φάρμακα σε περιοχές μακριά από την κατοικία τους. Προτιμούν λοιπόν το φαρμακείο της γειτονιάς τους. Έχουν δυσκολία να οδηγήσουν, να πάρουν το λεωφορείο, να στέκονται όρθιοι για πάνω από ένα τέταρτο κτλ. Αυτό είναι ο πρώτο λόγο. Δεύτερον, ε, χρειαζόμαστε τι συμβουλέ ε, του επαγγελματία φαρμακοποιού για τι παρενέργειε των φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε. Αυτό δεν γίνεται συνήθως από τον, συγκεκριμένο, από τον ειδικευμένο γιατρό, γιατί στο γιατρό πηγαίνουμε συνήθως δύο-τρει φορέ το χρόνο, ενώ ο γενικό παθολόγος που μπορεί να μα βοηθήσει έχει πάρα πολύ φορτό εργασία. Τρίτον, ο φαρμακοποιός που μα γνωρίζει και ξέρει ποια είναι ακριβώ η παθεσή μα μπορεί να μα δώσει συγκεκριμένε συμβουλέ και αν έχουμε συγκεκριμένε, παραδείγματο χάρη, ε, μολύνσει που μπορεί να προκληθούν, όπω παραδείγματο χάρη γυναικολογικέ, τα μάτια και αλλού και πριν να πάει κάποιος στο νοσοκομείο χρειάζεται να λάβει ε, κάποια επίγουσα περίθαλψη και επίσης πρέπει να δίνονται συμβουλές ε, για διάφορες θεραπείες που λαμβάνουμε για το πώς απαντά το νοσοποιητικό μας σύστημα στα κορτιζονούχα φάρμακα και πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δίνονται αυτές οι συμβουλές ε, προκειμένου να αποφεύγονται οι μολύνσεις και να αποφεύγεται μία επιπρόσθετη επίσκεψη στο γιατρό. Τέταρτον, εμείς αναμένουμε να μας συμβουλεύουν οι φαρμακοποίητες να μας λένε ποιες είναι οι άμεσες παρενέργειες και να μας ε, χορηγούν συγκεκριμένες συμβουλές. Σας ευχαριστώ κυρία Τέμπορα Φίλκης. Ε, με συγχωρείτε, σας παρακαλώ κύριε, μπορείτε να κάτσετε. Μπορείτε να κάτσετε κύριε, σας παρακαλώ. Salut. Sorry, can you sit down? Proszę bardzo, pani Debora Wilki. Με συγχωρείτε παρακαλώ, η κυρία Ντέμπορα Βέλκε. Καλημέρα σας. Εκπροσωπώ του ε, Βρετανού που κατεβούν ε, στην ε, περιοχή αυτή και εγώ είμαι υπέρ τους, του μεσογειακού συστήματο για την φαρμακευτική περίλαψη. Μόνο αυτές οι ειδικευμένε επιχειρήσει ξέρουν τους ε, πελάτες στην οικογενειακή ιστορία, ιατρική της ε, κλπ. Εάν υπάρχει αυτό το σύστημα που προτείνεται, θα εξαλειφθεί αυτή η ποιότητα. Το χειρότερα μάλιστα στην Υπεθρό ε, που δεν θα υπάρχει δυνατότητα κέρδους, θα εξαλειφθούν τελείως τα φαρμακεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα Ηνωμένη βρίσκεται, βρίσκονται συχνά τα φαρμακεία σε κέντρα εμπορικά, δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή στην οποία ζουν. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στο προσωπικό και δεν υπάρχει καμία σχέση με τους καταναλωτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ του ε, φαρμακοποιού και του ε, ασθενούς. Εμείς ε, σε περίπτωση καρκίνου είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με το φαρμακοποιό μας που ήταν στη θέση μας 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Δεν υπάρχει βέβαια τιμή γι' αυτό, αλλά οι πολυεθνικές βλέπετε ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Σας παρακαλώ, το μεσογειακό αυτό σύστημα ε, λειτουργεί πάρα πολύ καλά και μην το καταστρέψετε. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε. Σας ευχαριστώ. Τερέσα Βάρτη Χιβέντες έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Την ε, Επιτροπή. Λέγομαι Τέρσα Μαρτίν Χιμένες, είμαι φαρμακοποιός ε, και έχω, είμαι κάτοχος ιδιοκτήτρια φαρμακείου στο Τερεμολίνος. Εγώ έρχομαι εδώ για να περασπίσω ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να σχεδιάσει πόσο θεωρεί καλύτερο ότι πρέπει να γίνεται η παροχή φαρμακολογικών υπηρεσιών προκειμένου να προστατεύει τη δημόσια υγεία και το πώς θα πετύχει το στόχο αυτό. Βασίζομαι στο άρθρο 152, παράγραφος 5 της Συνθήκης της Ένωσης, όπως γνωρίζετε, ε, λέει ότι η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας είναι πλήρης αρμοδιότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους και αυτό αφορά την οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσίες Η Ένωση δεν έχει ε, μία πλήρη αρμοδιότητα για το θέμα αυτό της δημόσιας υγείας. Το φαρμακείο είναι ε, μία εγκατάσταση υπάρξει υγειονομική, υγειονομικό κέντρο δημόσιου συμφέροντος που ε, ουσιαστικά εξυπηρετεί τον πολίτη, το μοντέλο ε, που ρυθμίζεται, μάλλον το ρυθμισμένο μοντέλο που έχουμε στην Ισπανία μας βοηθά όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση. Οι φαρμακολογικές υπηρεσίες πρέπει να ασκούνται από τους επαγγελματίες φαρμακοποιούς. Εμείς έχουμε καταρτιστεί ακριβώς για το σκοπό αυτό και κόβεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας και παρέχουμε ποιοτική υπηρεσία στους πολίτες. Ε, έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ότι κάθε κράτος μέλος ε, είναι αρμόδιο για να σχεδιάζει το δικό του σύστημα υγείας και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία θα έπρεπε ε, να εξαρτώνται από τη Γενική Διεύθυνση της, την Γενική Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Υγείας Επίσης, ε, ο ε, φαρμακοποιός ε, θα πρέπει να συμμετέχει ο ίδιος στη χάραξη της υγειονομικής πολιτικής. Εμείς θέλουμε να παρέχουμε αξιόλογες υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια και εμείς ε, αυτό που κάνουμε, η φαρμακοποίηση είναι το εξή. Εγγυόμαστε την ανεξαρτησία μας, την επαγγελματική και την αμεροληψία μας στη χορήγηση των φαρμάκων. Συνεχίζουμε να είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες ε, και δεν ε, εξυπηρετούμε εμπορικά συμφέροντα. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών που να έχει ένα ελεύθερο και λογικό σύστημα υγείας που να διασφαλίζει την υγεία των ε, πολιτών, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Έτσι όπως ε, έχει το σύστημα στην Ισπανία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Γιατί να το ελέγξουμε. Εμείς θεωρούμε ότι το σύστημα της Ισπανίας λοιπόν θεωρεί πολύ καλά. Κυρία Μπεγκόνια Πέρας, δύο λεπτά. Καλημέρα σας. Ε, για να ε, μην ε, αναγνω... εδώ σας ζητάμε να μην ε, αναγνωρίσετε το ότι είναι παράνομα ο τρόπος που λειτουργούν τα φαρμακεία της Ισπανίας. εδώ, ο, μάλλον το 1974 ο Φράνκο είχε θέσει αυτούς τους περιορισμούς και από τότε οι διάφορες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αυτούς τους περιορισμούς για να ωφελήσουν τους εγκατεστημένους ήδη φαρμακοποιούς και υπάρχει έτσι ένα σύστημα τιμών στο οποίο παρεμβαίνει το κράτος, ο οποίος είναι ο κύριος πελάτης. Αυτό δεν έχει να κάνει με κανένα ανάλογο προστασίας της υγεία. Ε, το κράτος εδώ ουσιαστικά θέτει κανόνες που να εμποδίζουν το να ανοίξουν νέα φαρμακεία. η ε, πλαφάρμα δεν θέλει μία απορρίθμιση αλλά αύξηση του ελέγχου της ε, δίκησης ε, των φαρμακείων σε ένα σύστημα ανοιχτά ελεύθερο. Υπάρχουν οι εξής λόγοι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος υγειονομικός λόγος που να αιτιολογεί τον περιορισμό του ελεύθερου ανοίγματος και δεύτερος είναι ότι είναι άδικο να εμποδίζουμε σε Ευρωπαίους φαρμακοποιούς να ασκήσουν ελεύθερο το επάγγελμά τους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι το κατάλληλο για να εγγυηθούμε την ορθή παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Υπερασπιζόμαστε ότι η απελευθέρωση θα επιφέρει μεγαλύτερη ποιότητα στη χορήγηση των υπηρεσιών. Είναι ε, προφανές ότι ο περιορισμός ε, τελικά περιορίζει την πρόσβαση του πολίτη στην παροχή φαρμάκων. Ε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Δύο λεπτά. Κύριε Μοράλες. Buenos días. Καλημέρα σα. Το 1994 ζήτησα, να ανοίξω ένα φαρμακείο στο Τερέρο, ε, στο Νταϊμένο, όπου εκεί ε, πραγματικά ήταν, είχαμε πάρα πολύ λίγα φαρμακεία, είχαμε μόνο 7 και τότε εγώ ουσιαστικά σεβάστηκα την υφιστάμενη νομοθεσία το εν λόγω διάταγμα στο οποίο βασίστηκα επέτρεπε να ιδρυθεί ένα φαρμακείο πάντοτε αν υπήρχε πληθυσμός άνω των 2.000 κατοίκων και το πιο, μακρινό, το πιο κοντινό φαρμακείο να βρίσκεται 500 μέτρα μακριά. Ε, οι γείτονε είχαν ε, επισημάνει στο Δήμαρχο ότι χρειαζόταν να ανοίξει στη γειτονιά αυτή ένα συγκεκριμένο φαρμακείο. Εγώ ζήτησα ε, από το Δήμο την άδεια και μου αρνήθηκαν. Το ζήτησα και από το Δήμο της Ματρίτης και επίσης μου αρνήθηκαν. Και ε, τότε προσέφυγα στο δικαστήριο. Τέσσερα χρόνια μετά, το Μάιο του 1998, το Δικαστήριο της Καστίγια Λαμάντσα αποφασίζει ότι επιτρέπεται το να ανοίξει ένα φαρμακείο στο Τερέρο, στο Νταϊμιέν και λέει αυτή η απόφαση ότι ε, πρέπει να, υπάρχει, να ληφθεί υπόψη καταρχήν η υπηρεσία, η δημόσια που θα χορηγήσει αυτό το νέο φαρμακείο στην περιοχή. Επίσης, ε, ε, μάλλον υπήρχε προσφυγή αυτής της απόφασης από τους ανταγωνιστές και το 1999 υπήρξε αποτέλεσμα. Εγώ τελικά προσωπικά έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Οι γείτονε ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τι υπηρεσίε. Το 2003 αποφάνθηκε το ανώτατο δικαστήριο τη Μαδρίτη και ανέστηλε, ανακάλεσε την προηγούμενη απόφαση και είπε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη γειτονιά δεν υπάρχει δυσκολία από του γείτονε να πάνε πιο μακριά για να αγοράσουν τα φάρμακά του. Αυτό εγώ δεν ε, το κατανόησα αυτή την απόφαση. Έτσι λοιπόν ε, κλείνει στη συνέχεια ε, το φαρμακείο και οι άλλοι φαρμακοποιοί μου ζητούν να τους δώσω 11 εκατομμύρια πεσέτες που έπρεπε να δώσω τότε στους φαρμακοποιούς για απώλεια, για ζημία. Όμως ε, οι γείτονες ήλθαν για να υπερασπίσουν, να αποτρέψουν το να κλείσει το φαρμακείο και μάλιστα χρειάστηκε να παρέμβει και η αστυνομία. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν πρόκειται να ολοκληρώσουμε σήμερα την εξέταση της αναφοράς της προφανώς. Θα ήθελα όμως τώρα να παρακαλώ στην Κομισιόν να τοποθετηθεί επί του θέματος. Δύο λεπτά κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σύντομα ποια είναι η κατάσταση. Αρχίσαμε διαδικασία παραβίας, παράβασης και το 2006 υπήρξε ένα πρώτο βούλευμα και υπευλήθησαν δύο περιορισμοί. Πρώτον στην ιδιοκτησία, δεύτερον στην τοποθεσία. Και καταλήξαμε ότι οι περιορισμοί αυτοί τελικά δεν εξυπηρετούν στόχους δημοσίας υγείας. Δεν έχουν καμία σχέση. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι δεν συμφωνούν με το άρθρο 43 της συνθήκης που προβλέπει την ελεύθερη εγκατάσταση επιχειρήσεων. Συμμεριζόμαστε πλήρως την ανησυχία σας για την προσβασιμότητα που είπατε και γι' αυτό ακριβώς αρχίσαμε μια πολύπλευρη συζήτηση με ενδιαφερόμενους για αυτά τα θέματα. Τον Οκτώβριο έγινε ένα σεμινάριο για την προσβασιμότητα γεωργικών υπηρεσιών και επίσης έχουμε επικοδομητικούς διαλόγους με την Ισπανική κυβέρνηση παράλληλα με τις διαδικασίες για παράβαση πρόσφυγες. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα μας για τα συμπεράσματα του σεμιναρίου εκείνου, αλλά ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς το θέμα και της τοποθεσίας και της πρόσβασης που υπάρχει ή δεν υπάρχει σε γεωργικές υπηρεσίες, σε φαρμακευτικές υπηρεσίες. Ζητήσαμε πληροφορίες από τις οργανώσεις φαρμακοποιών και τα στοιχεία που μας έδωσαν τα αναλύουμε τώρα και θα οργανώσουμε και δεύτερο σεμινάριο τον Ιούνιο. Αν υπάρχουν απορίες να τις λύσω. Κυρίες και κύριοι, έχω πέντε ακόμη ομιλητές και ομιλήτριες. Ένα λεπτό ο καθένας. Αλλά παρακαλώ τους βουλευτές επίσης να προτείνουν κάποια λύση. Δεν θέλω γενικές τοποθετήσεις, αλλά προτάσεις. Τι να κάνουμε. Πάντως δεν θα λήξει σήμερα η υπόθεση. Παρακαλώ όμως να μας κάνετε και προτάσεις. Κύριος Τζάπαλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει όσο είπε η Κομισιόν, Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επιπραβάση το 2001. Δεν ήταν επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Υπόθηκε αυτό και νομίζω ότι θα ήταν καλό να δούμε αν υπάρχει επικαιροποίηση των στοιχείων. Ε, η περίπτωση ε, που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα πραγματικά είναι κατά του Ευρωπαϊκό δικαίου, κατά τις οδηγίες για τα προσόντα, για τα επαγγελματικά προσόντα, κατά τις οδηγίες για την απελευθέρωση των περισσιών ε, Έτσι λοιπόν, αν η Κομισιόν εμβαθύνει επί του θέματος και ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ναι, εγώ καταρχήν πιστεύω Καταρχήν ε, θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να αποσύρεται αυτή τη διαδικασία υπερβάση γιατί η Κομισιόν μας είπε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να διερευνήσει. Δηλαδή καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσετε την υπόθεση και μετά να δείτε αν ξεκινάτε διαδικασία υπερβάση γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για την απελευθέρωση μιας αγοράς αλλά μιλάμε για ένα θέμα που πηγαίνει πολύ πιο πέρα μιλάμε για τη δημόσια υγεία έτσι λοιπόν πρέπει πραγματικά να διερευνήσουμε το θέμα εις βάθος και ε, στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει παράβαση, τότε να ξεκινήσετε διαδικασία επί παραβάση. Ε, εγώ προέρχομαι από την Αβάρα και θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιό να κάνει μια μελέτη για το τι έγινε το 2003 όταν είχαμε ψευδοαπελευθέρωση, όχι απόλυτη απελευθέρωση γιατί άνοιξαν εκεί κάποια φαρμακεία αλλά και άλλα έκλεισαν και τελικά ε, δεν υπήρχε αύξηση των υπηρεσιών ε, της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στους πολίτες. Ευχαριστώ. Τουργάι. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με το συνάδελφο. Νομίζω ότι το πρώτο που ζητά δημόσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι να ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Δεν ξέρω εδώ, ε, ε, στην Ισπανία παρέχεται, διασφαλίζεται μία καλή παροχή υπηρεσιών και καθώς εδώ μας δίνεται πάρα πολύ λίγο χρόνο, εγώ θέλω να ζητήσω και το εξή. Εδώ δεν έχουμε μία επιτροπή υγείας, αλλά έχουμε μία επιτροπή εσωτερικής αγοράς. Ίσως αυτή η επιτροπή και η επιτροπή αναφορών θα έπρεπε να γράψει στον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς να μελετήσει αυτό το πρόβλημα και να συζητηθεί και το θέμα αυτό σε εκείνη την επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκουτιέρες. Ένα λεπτό. Εγώ νομίζω ότι κατανοείται ορισμένες από τις αναφορές και πραγματικά με εκπλήσει η περίπτωση ε, που δείχνει την αδικία περίπτωση της κυρίας Δεν ξέρω, συμφωνώ εγώ Νομίζω ότι η απελευθέρωση δεν είναι η λύση. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί φαρμακοποιοί εξαπατήθηκαν ε, γιατί πίσω από την απελευθέρωση βρίσκονται μόνο οι μεγάλες εταιρείες και τελικά αντί να έχει κάποιος ένα φαρμακείο απλώ θα γίνει υπάλληλο μια μεγάλη εταιρεία. Εγώ πάρα πολλά χρόνια δίνω αυτή τη μάχη και βλέπουμε έχουμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ούτε καν ισπανικές που είναι κατά του υφιστάμενου συστήματος. Εγώ νομίζω ε, ότι δεν πρέπει να εξαρτώνται ε, τα φαρμακεία από το προϊόν που πουλάνε, αλλά από την υπηρεσία που παρέχουν. Μιλάμε για μια υγειονομική υπηρεσία. Δεν μπορούν λοιπόν να καλύπτονται από την οδηγία υπηρεσιών. Ε, επίσης, Νομίζω ότι εδώ πραγματικά παίζουμε με το θέμα της υγείας. Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να πω προσοχή γιατί τελικά σας εξαπατούν. Γιατί θα καταντήσετε να είστε υπάλληλοι μεγάλων πολυεθνικών. Και κοιτάξτε, ξέρουμε τι έγινε και με την περίπτωση του Καρφούρ. Pan Angela ένα ένα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα να μιλήσω γιατί είμαι φαρμακοποιός δεν έχω ανοίξει ποτέ φαρμακείο, δούλεψα στη βιομηχανία. Θεωρώ ότι η απελευθέρωση του επαγγέλματο στην Ισπανία προσυδειάζει με τι τάσει που υπάρχουν στη χώρα μου, την Ελλάδα. Θεωρώ ότι όλη η ιστορία είναι γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώ. Η παρουσία φαρμακοποιού στο φαρμακείο εξασφαλίζει πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων οικονομίε και στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, με τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγεία. Αλλά θέλω να κλείσω λέγοντα το εξή. Σε ερώτησή μου προ τον Επίτροπο Μακρύ πριν από τρεις μήνες, μου απαντήθηκε επισήμως ότι μέσα στο 2009 θα γίνει μια διαβούλευση όπου κάθε χώρα μέλος θα στοιχειοθετήσει για ποιους λόγους έχει περιοριστικά μέτρα στο επάγγελμα. Γιατί δεν περιμένει η Επιτροπή να τελειώσει αυτή η διαβούλευση και να δούμε πού, πού πηγαίνει. Αυτό ήθελα. Proszę Państwa, więc tutaj ze wszystkich wypowiedzi... ευχαριστώ. Όλοι το λόγο σήμερα. μα ε, ότι δεν ε, πρόκειται να κλείσουμε την αναφορά σήμερα. Προφανώς δεν μίλησαν όλοι ενεφέροντος ακριβώς πάνω στο ίδιο θέμα. Από όσα ακούσαμε όμως από τους δικούς μας βουλευτές, παραδείγματος χάρη τους βουλευτές, μα οδηγούν να καταλήξουμε στα εξή συμπεράσματα. Απελευθέρωση αυτής τη συγκεκριμένη αγορά ίσω είναι επικίνδυνη, γιατί πράγματι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί κανένα να ελπίζει απλώ ότι θα επιληθούν τα προβλήματα όταν περάσουμε σε μεγαλοβιομηχανίες και νομίζω ότι προ όφελο των καταναλωτών και των πολιτών είναι καλύτερο να υπάρχει ένα φαρμακείο της γειτονιάς. Είναι σαφές νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Και υπάρχει μια σειρά ε, δυνάμει ψηφισμάτων εδώ και θα παράσουμε νομίζω στην Επιτροπή ΕΜΚΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Και πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει δική σας άποψη. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να καταπολεμηθούν προσπάθειες για την εισαγωγή μονοπωλίου. Θα διατηρήσουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά αυτή και όπως σας είπα θα έρθουμε σε επαφή με την Κομισιόν και την αρμόδια επιτροπή να δούμε τι θα κάνουμε. Ένα λεπτό κύριε Γουτιέρης. Ένα λεπτό. Θέλω να σας πω ότι ε, ε, ε ότι υπάρχει Επιτροπή για την Υγεία και εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να συζητηθεί όπου συζητήσαμε και το θέμα της κινητικότητας των ασθενών. Ωραία, θα το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε σίγουρα. Θα έρθουμε σε επαφή με την εποχή ΙΜΚΟ και την ε, ε Επιτροπή για το θέμα αυτό. Και θα συνεχίσουμε μετά τις συζητήσεις. Ωραία. Ελπίζω πράγματι ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση που θα είναι υπέρ της άποψής σας. Πέρα συνεδρίωση αυτή θα τα ξαναπούμε στις 3.